sur l'échange de vues avec la Commission. D'accord. Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ πολύ. Άρχε τη συνεδρίαση. Αν δεν έχετε παρατηρήσει, θεωρώ εγκεκριμένη την ημερήσια διάταξη. Οι αποφάσεις των συντονιστών της 28ης Ιουνίου βρίσκονται ε, στο φάκελο τα έγγραφά σας και αν δεν έχετε αντιρρήσεις από πλευρά σας θεωρώ ότι εγκρίνεται το σύνολο των πρακτικών. Έχετε και τα πρακτικά μπροστά σας των προηγούμενων συνεδριάσεων από την πλευρά της Διευμηνίας να θυμίσουμε ότι είναι η 36η ημέρα κινητοποιήσεων, η διοίκηση εξακολουθεί να μην δείχνει πνεύμα συνεργασίας, γι' αυτό συνεχίζουμε και γι' αυτό ακριβώς με τα λύπη μας σας ενημερώνουμε ότι θα διακόψουμε ακριβώς με το τέλος της προβλεπόμενης διάρκειας. Συνεχίζει, ο πρόεδρος, με την κτηριακή ε, πολιτική του Κοινοβουλίου. Έχω εδώ τον, τους αντιπροέδρους Σασόλη και Βίλαντ, όπως και το Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βέλε, τους καλωσορίζω. Στόχος αυτής εδώ της συνεδρίασης είναι να συλλέξουμε σημαντικές πληροφορίες στον τομέα της κτηριακής πολιτικής του Κοινοβουλίου και ε, σχετικά με τις συνέπειες σε επίπεδο δημοσιονομικό. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών βασίζεται στο ετήσιμο έγγραφο εργασίας για την κτηριακή πολιτική, το οποίο για το 18 το λάβαμε στο τέλος Μαΐου, όπως επίσης και στο έγγραφο στρατηγική κτηριακή μετά το 19 που πήραμε πρόσφατα. θα έχουμε κάποιες ε, ενδείξεις και για το μέλλον του κτηρίου PHS. Ε, δεν θα σας καθυστερήσω άλλο, λέει ο Πρόεδρος, και θα δώσω το λόγο 8 με 10 λεπτά στον κάθε ένα από τους ομιλητές. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο Αντιπρόεδρος κ. Βίλαντα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν θα εξαντλήσω εντελώς και τα 8 λεπτά. Επιγραμματικά μόνο, να πω μερικά πράγματα. Σε τελευταία συνεδρία του Προεδρείου, πιστεύω, μιλήσαμε για την κτηριακή πολιτική, που είναι μακράς πνοή σχέδια. Και στο κτίριο PHS προχωρήσαμε ένα βήμα. Αποφασίσαμε βάσει μελέτης ε, σκοπιμότητας να ελέγξουμε αν υπάρχει δυνατότητα ανακαίνησης, ενίσχυσης στην ασφάλεια και βελτίωσης από τη μια ή από την άλλη εάν χρειάζεται αναδιάρθρωση, δηλαδή να χτίσουμε καινούριο κτίριο. Αν είναι καλύτερη αυτή η λύση. Δεν αποφασίσαμε καμία από τις δύο ε, λύσεις. Ε, απορρίψαμε και διατήρηση του status quo και γενικός γραμματέας ε, στην αρμόδια ομάδα εργασίας για τα κτίρια εξήγησε τη φάση στην οποία βρισκόμαστε για μια πιο ενδελεχή βολιδοσκόπηση για να πάρει μια απόφαση το Προεδρείο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Έτσι κι αλλιώς θα χρειαζόταν αυτή η φάση τώρα. Δηλαδή δεν χάνουμε επιπλέον χρόνο, τον οποίο έχουμε χάσει ήδη στο παρελθόν. Δεν θα το αντικρούσω. Ε, θα προτιμούσα πριν από δύο χρόνια να βρισκόμασταν εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Επίσης ε, θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε το εξής. Ανεξάρτητα τώρα από την ανακαίνιση και τις εργασίες που θα γίνουν και ανεξάρτητα από την ε, αναδιάρθρωση ή την ανέγερση νέου κτίριου ε, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το ευρύτερο περιβάλλον έχουν προκύψει νέες εξελίξεις. Είμαστε σε επαφή με το Δήμο των Βρυξελών και για να έχουμε αποδοχή στον κόσμο και στη γειτονιά ε, θα πρέπει να φροντίσουμε ε, σε αυτό το οικόπεδο που είναι το τρίγωνο των Βερμούδων ουσιαστικά ανάμεσα στα τρία ε, θεσμικά όργανα ε, ε, και μεταξύ αυτών και το πάρκο Λεοπόλτ ε, να υπάρχει ένα συνδυασμό αστικής περιοχής, τουριστικών ενδιαφερόντων και άλλων δραστηριοτήτων. Γιατί είναι και ένα σχολείο εκεί. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν υγιές μείγμα που να συνδυάζει την, ημερινή, την ημερήσια δραστηριότητα, συγγνώμη, την βραδινή δραστηριότητα και το Σαββατοκύριακο. Έτσι θα αυξηθεί και η αποδοχή του κοινού ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, το καθεστώς ασφαλείας του κτηρίου PHS. Θα παρακαλούσα όλα τα μέλη της Επιτροπής Προπολογισμών να μεταβούν στο αναγνωστήριο για να διαβάσουν όλα τα έγγραφα που δεν είναι δημόσια και δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ξέρω ότι ε, ο κύριος Μάνκα, ε, ο οποίος είναι και μηχανικός, έχει δει τα έγγραφα αυτά. Καλό θα ήταν οι πολιτικές ομάδες να ορίσουν ένα συνάδελφο ο οποίος θα τα παρακολουθεί και θα πάει να διαβάσει τα έγγραφα αυτά για να γνωρίζει περί τίνος πρόκειται και να ξέρουμε πώς έχει η κατάσταση έτσι, σε μεγαλύτερο βάθος. Για το κτίριο Μάρτενς ε, άρχισε να λειτουργεί. Εγώ το είχα επισκεφτεί και ως εργοτάξιο. Ε, αφού του παραδόθηκε πρέπει να πω ότι είναι πολύ υψηλή αξία του και έχω την εντύπωση ότι πέτυχε κιόλα. Πολύ ωραίο κτίριο. Έχετε τη δυνατότητα να πάτε και να φάτε εκεί στο εστιατόριο για να ε, αποκομίσετε και ιδία άποψη. Οι υπάλληλοι που εργάζονται εκεί είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι για το κτίριο μου του ΑΓΕ. είναι ε, το κτίριο με τις αίθουσες σεμιναρίων και μαθημάτων. Πάει καλά το εργοτάξιο και θα τελειώσει μάλλον και νωρίτερα από ό,τι έχει προβλεφθεί. Στα κράτη-μέλη τώρα. Ακούσαμε ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα ως προς τη χρηματοδότηση και μάλιστα ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ε, ομάδα εργασίας Brexit του Προεδρείου, νεοσύστατη είναι αυτή, θα συζητήσουμε τις επιπτώσεις του Brexit και για το Κοινοβούλιο θα συζητήσουμε και τα θέματα του Λονδίνου και του Εδιμβουργού και τα δύο κτίρια είναι μισθωμένα και υπάρχουν ε, διάφορα σενάρια. Θέλουμε να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Ακόμα απέχουμε πολύ από μια απόφαση. Ε, είναι νωρίς. Γενικά θέλω να πω το εξής. αρμόδιος επίτροπος είναι ο κύριος Σέτιγκερ και με τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή Επικοινωνία ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχω συζητήσει και με τους δύο. Δεν μ' αρέσει το γεγονό ότι δεν επικρατεί παντού έτσι μια αγαστή συνεργασία και ωραία ατμόσφαιρα συνεργασίας. Από όλα έχει ο Μπαχτσές ε, Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή πηγαίνουν σε μια πρωτεύουσα και θέλουν να αγοράσουν ένα κτίριο. Τις παραμονές της αγοράς ε, βγαίνει η Κομισιόν και λέει «Α, δεν θέλω να αγοράσω, θέλω να νοικιάσω». Στο Παρίσι χάσαμε εκατομμύρια γιατί δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε για το κτίριο, διότι η Κομισιόν τα στείλωσε κυριολεκτικά. Και τα ε, το, τα έξοδα, ούτε τα μοιραζόμαστε δίκαια για τα τετραγωνικά που μισθώνουμε, ε, ούτε υπάρχει καλή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω από το 2019 και μετά να αλλάξει αυτό. Για παράδειγμα, και θέλω να το πω ξεκάθαρα. Είναι συνήθιστο το ένα όργανο να χρεώνει τόκους στο άλλο, αλλά όταν σου λέει ένα όργανο εγώ δεν αγοράζω και πήγαινε εσύ κοινοβούλιο να αγοράσεις το κτίριο, Μέχρι και μια πενταετία αργότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μισθώνει το κτίριο και για μένα είναι προφανές ότι θα πρέπει να καταβάλει και το ε, αντίστοιχο ενίκιο όταν δεν είναι ιδιοκτήτης και είμαστε εμείς. Δεν ξέρω μήπως χρειάζεται κάποια συμφωνία έτσι Τέλος θέλω να πω ότι κάναμε μια πιλωτική φάση τώρα. Ε, προκήρυξαμε ένα διαγωνισμό για τα, ε, τα έπιπλα, για τον εξοπλισμό και πάλι δεν ξέρουμε αν θα τα αγοράσουμε, αν θα τα νοικιάσουμε. Πέντε είναι οι κατασκευαστές ε, που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Και πρόκειται για τρεις χώρους. Είναι ένα γραφείο με πλήρη εξοπλισμό, ένα γραφείο χωρίς εξοπλισμό και ένας χώρος αναμονής. Ε, αρμόδιοι ε, είναι η κυρία Μωρέ Σαρτιέ, που έχει η κυρία Μωρέ Σαρτιέ ήδη ένα πιλωτικό <coughs> γραφείο, η κυρία Κέπχαρτ, η κυρία Χάουταλα, ο κύριος ε, Σασόλη και ο υποφαινόμενος. Ελάτε να τα δείτε τα γραφεία αυτά. Έχουμε ε, πολύ τεχνογνωσία και για τον τρόπο λειτουργίας ε, του γραφείου και έχουμε αποκομίσει και πολλές ε, εμπειρίες και εντυπώσει. Είναι πιο ευέλικτη αυτή η μορφή λειτουργίας του γραφείου και στο μέλλον θα μας βγει και φτηνότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα επανέλθουμε στο θέμα της ενίσχυσης των σχέσεων ανάμεσα στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Ο κύριος Σασόλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπε και ο συνάδελφος Βίλαντ, ε, υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να ε, θέσουμε. Με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, με την αλλαγή της θεσμικής αρχιτεκτονικής που ακολούθησε τη συνθήκη της Λισαβόνας, προκλήθηκαν και θα προκληθούν επίσης περαιτέρω συνέπειες της δραστηριότητες του Κοινοβουλίου. Σκεφτείτε ότι μετά τη Λισαβόνα αυξήθηκαν οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου όπως και οι ευθύνες του και η αποστολή του και αυτό επηρεάζει ακριβώς και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμεθα τα κτίρια. Ε, για το τέλος του 2018 έχουμε οργανώσει 800 περίπου τριγωνικούς διαλόγους. Καταλαβαίνετε πόσο περίπλοκο είναι, ε, αλλά έχουμε μόνο τέσσερις αίθουσες για να το κάνουμε αυτό σαν κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε την θεσμική αρχιτεκτονική με την δυνατότητα χωροτακτικά του Κοινοβουλίου να ανταποκριθεί. Ναι, απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να καταστεί ικανό να λειτουργήσει με τον ευρυθμότερο τρόπο. Το λέγω αυτό γιατί πολλές από τις ε, προτάσεις και παρουσιάσεις που έγιναν για την, τον εξυγχρονισμό ακριβώς των κτηριακών εγκαταστάσεων οφείλονται και προέρχονται από τις αλλαγές ε, του ρόλου και της δραστηριότητας. Έχουμε δηλαδή και πρέπει να έχουμε μια κτηριακή πολιτική που να ακολουθεί τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου. Τώρα για το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Αντιπρόεδρος Βίλαντ, να πω ότι στις Βρυξέλλες ε, με την έναρξη δραστηριότητας του κτηρίου του κτηρίου Μέρτενς όπως επίσης και του νέου κτηρίου ε, του πρόσφατου κτηρίου στο, ε, στην πλατεία Ντεμεούς μπορούμε να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας όχι απλά κατάλληλες αλλά εξαιρετικές συνθήκες εργασίας. Στο Στρασβούργο ε, τίθεται το ίδιο περίπου θέμα με το κτίριο Άβελ το οποίο λειτουργεί πλέον από το 17 μας δίδεται η δυνατότητα να προσφέρουμε στους ε, ε, ευρωβουλευτές μας μια πλέον κατάλληλη χωρική αν θέλετε ένα χωρικό περιβάλλον. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει χώρο στο Στρασβούργο, δεν υπάρχει ιδιωτικότητα. Αν θέλετε να κάνετε ένα εμπιστευτικό τηλεφώνημα που ζητάτε από τους συνεργάτες σας να βγούνε από το από, την, από το χώρο, από το γραφείο. Οπότε τώρα με τον δεύτερο χώρο θα μπορέσουμε να εργαστούμε με πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. σχετικά με τώρα με το παρλαμεντάριο, τα παρλαμεντάριο. Ε, όλα έχουν στεφθεί από επιτυχία. Οι Βρυξέλλες είναι το δεύτερο σημείο το οποίο επισκέπτεται ο κόσμος μετά από την Grand Place. Και στο Στρασβούργο είχαμε περισσότερους ε, επισκέπτες από ό,τι περιμέναμε. Το ίδιο συμβαίνει και στο Βερολίνο και στη Λιουμπλάνα. Επίσης είναι πολύ καλή πρωτοβουλία για την έκτακτη παρουσία των παρλαμεντάρι ε, στα διάφορα, στις διάφορες ε, πρωτεύουσες και χώρες κάτι το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί, αν θέλετε, μια παιδαγωγική ευρωπαϊκή δραστηριότητα. Σχετικά τώρα με την ανακαίνιση των χώρων της ε, αναδιαρρυθμίσεις και την ασφάλεια. Λοιπόν, θα πρέπει να συνεχίσει η προσπάθεια να καθίστανται τα κτίρια του Κοινοβουλίου ασφαλέστερα, αυτό είναι σαφές, ιδιαίτερα μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν το 2015 και 2016. Αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα. Ξεκινήσαμε λοιπόν την προσπάθεια αναδιάφρωσης και αναδιαρρύθμισης των συνθήκων ασφάλειας και αυτή η προσπάθεια μας επιτρέπει σήμερα να ε, έχουμε βελτιώσει την αξιολόγηση των κινδύνων τους οποίους αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα. Προγραμματίσαμε επίσης και ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων ε, σταδιακά για τα επόμενα χρόνια για να γίνουν ασφαλή και τα υπόλοιπα κτίρια του Κοινοβουλίου γιατί δεν έχουμε μόνο τις κεντρικές εισόδους, έχουμε πάρα πολλά κτίρια και όλα φυσικά θα πρέπει να γίνουν ασφαλέστερα. Τώρα, για τα κτίρια που έχουμε στην διοκτησίες μας. Ξέρετε ότι τα κτίρια τα οποία ανήκουν στο δημόσιο τομέα έχουν μια ισχυρή παρουσία, αν θέλετε. Φαίνονται Συνεπώς εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμεθα τους κανόνες που επιβάλλουμε στους άλλους, διότι εμείς αποφασίζουμε για πολλά, κάνουμε πολλούς νόμους και είμαστε οι πρώτοι πολλές φορές που δεν τους σεβόμεθα. Αναφέρομαι λοιπόν στην οδηγία του 2012-27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα. Εμείς συζητάμε σε σχέση με αυτή την οδηγία από τους άλλους να την σέβονται, οπότε πρέπει να δώσουμε το σωστό παράδειγμα. Επιβάλλει η οδηγία αυτή το 3% των καλυπτόμενων χρήσιμων επιφανειών που ψύχονται ή θερμαίνονται, ιδιόκτητες επιφάνειες, θα πρέπει σε αιτήσια βάση να ελέγχονται έτσι ώστε να γίνονται σεβαστά τα κατώτερα αποδεκτά επίπεδα αποδοτικότητας. Όταν βάλουμε ε, λοιπόν το 3% του συνολικού χώρου που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας, καταλήγουμε σε 36.000 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία θα πρέπει κάθε χρόνο να αλλάζουν και να ελέγχονται για τα επόμενα τρία χρόνια. Βλέποντας το σύνολο των κτηρίων που έχει ιδιόκτητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σημαίνει ότι κάθε κτίριο θα πρέπει να υποβάλλεται σε έναν έλεγχο και μια ουσιαστική αλλαγή κάθε 33 χρόνια. Μιας και πρόκειται για μια ευρωπαϊκή οδηγία, την οποία εμείς με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε να προωθήσουμε σχετικά με τα δημόσια κτίρια, Έχουμε λοιπόν και το ηθικό καθήκον να δώσουμε πλέον το σωστό παράδειγμα. Ευχαριστώ κύριε σας όλοι μου που μας υπονθυμίσατε τις υποχρεώσεις μας, τον σεβασμό των κανόνων που πρέπει πρώτοι να επιδείξουμε. Ο Γενικός Γραμματέας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε ότι μέσω της απόφασης του Προεδρείου τον προηγούμενους μήνες Έχουμε πετύχει κάτι πολύ καλό στην κτηρική πολιτική. Όσον αφορά την μεσοπρόθεσμη στρατηγική, είναι ξεκάθαρο ότι στο Στρασβούργο δεν έχουμε περισσότερη ε, ανάγκη για άλλα κτίρια, είτε να κατασκευάσουμε είτε να νοικιάσουμε στο Λουξεμβούργο. Παράλληλα με το project που τρέχει το να γίνει ενωπής των κτίριων δεν υπάρχει περαιτέρω ανάγκη χώρου και ότι στις Βρυξέλλες δεν είναι απαραίτητη η ενοικίση άλλων χώρων στο κέντρο όπως το παρελθόν αλλά έχουμε άλλες προτεραιότητες έχουμε για τις Βρυξέλλες το τρεύδιο, το κτίριο. Και υπάρχουν και τρεις προτεραιότητες του Προεδρείου. Πρώτον, χρειαζόμαστε περισσότερες δυνατότητες για τριμερή διάλογο, γιατί δεν ε, συμβαίνουν συχνά όσον αφορά την εκτηριακή πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν, ε, εν αυτό το χρόνο να αποφασίσει το Προεδρείο, πότε θα πρέπει να οργανώσουμε στους διαλόγους για το παρλαμεντάρια αναφερθήκατε σε όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δημιουργηθούν, να καθιερωθούν Έχουμε καλές εμπειρίες μέχρι στιγμής και τρίτον υπάρχει μια συστηματική πολιτική αναγέννηση, πρέπει να υπάρξει μια πολιτική αναγέννηση και υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2050 πότε και ποιο κτίριο θα πρέπει να αναγκαινιστεί για να αποπολιτοποιήσουμε τέτοιου είδους αποφάσεις. Αυτό που είπε και ο ε, αντιπρόεδρος Σασούλη, το 3% των κτηρίων πρέπει να ανακαινιστεί. Υπάρχει σαφήνεια προς αυτό και υπάρχει μια ξεκάθαρη αλλαγή ως προς την πολιτική του παρελθόντος. Κατά δεύτερον, το Προεδρείο μετά από πολλά χρόνια, ε, η πρώτη διαβούλευση έγινε το 2010, έλαβε μια απόφαση για την εξοικονόμηση για το κτίριο ΣΠΑΚ ενεργειακή ε, εξυγίαση και με μια νέα λειτουργία, ε, μια νέα κατασκευή με βάση ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες ε, του κάθε κόνσεπτ. Θα πρέπει να διαρκέσει 1,5 χρονό ε, αυτός ο διαγωνισμός μέχρι το τέλος του 2010 θα πρέπει να έχουμε μια πρόταση στο τραπέζι ώστε τον Ιανουάριο του 2020 ε, να ξεκινήσει ε, να ξεκινήσουν οικοδομικέ εργασίε. Κατά τρίτον, έχουμε το κτίριο Μάρτεν, στο οποίο άνοιξε τις πόρτες τους και έχετε τη δυνατότητα να το δείτε. Αν είναι ένα ποιοτικό άλμα σε σχέση με τα κτίρια που είχαμε μέχρι τώρα, ε, ε, ισχύει αυτό γιατί υπήρχε διαβούλευση με τους χρήστες ε, για την χρηστικότητά του και βλέπουμε επίσης τη θετική επίδραση που, που είχε ο διάλογος που έγινε New World on Work. Και βλέπουμε λοιπόν ότι βασίζεται όλο στο διάλογο την επικοινωνία ώστε να είναι προσαρμοσμένα τα κτίρια στις ανάγκες ε, των γενικών διευθύνσεων. Υπάρχει λιγότερος χώρος για τους ε, συνεργάτες, αλλά είναι διαφορετικά οργανωμένος ο χώρος. Η αντίδραση των συνεργατών ε, είναι θετική και αυτό το κτίριο θα αποτελέσει και το πρότυπο για το νέο κτίριο στο Λουξεμβούργο και για το κτίριο Μονταγέ συμμετοχή 63. Έχουμε ένα ποιοτικό άλμα ε, όσον αφορά την οργάνωση, η οποία θα δώσει πρόσβαση στο 50% των ε, συνεργατών. η αντιπρόεδρος επίσης είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Έχουμε ένα νομοθεσία στο Στρασβούργο για το ένα συν ένα. Θα πρέπει καθένας να έχει το να έχει το δικό του γραφείο και ένα ξεχωριστό γραφείο για τον βοηθό. Έχουμε τον εκτήριο Χάβελ, αλλά και η διοίκηση θα πρέπει να έχει τον χώρο, γιατί δεν είναι αποδεκτό πλέον οι ε, βουλευτές να έχουν το δικό τους γραφείο. Εδώ στη Βρυξέλλες έχουμε ένα με δύο για κάθε ε, βουλευτή. Μπορεί να έχει δύο γραφεία επιπλέον για κάθε συνεργάτη. ένα χώρο για να δέχεται κόσμο. Αυτός λοιπόν, αυτό το μισό έτος ήταν πολύ καλό και προχωρήσε σε μια νέα ποιότητα για την τελική πολιτική. Eh Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Θα ζητήσουμε τώρα από τον, την εισηγήτριά μας, την κυρία Χολμέιερ, να αξιολογήσει και αυτή την κυριακή μας πολιτική. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Γενικέ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ καταρχάς για την ανταλλαγή αυτή απόψε. Δεν θέλω να σας κρύψω ότι τους τελευταίους μήνες είχαμε κάποια προβλήματα στην πολιτική επικοινωνίας και το λέω έτσι ειλικρινά και ανοιχτά και παρακαλώ και το λέξω ονόματος όλων των συναδέλφων αυτό να έχουμε όλα τα έγγραφα. Έτσι ώστε πρώτα απ' όλα να μπορούν οι συνάδελφοι να τα διαβάζουν και δεύτερον να έχουν και ποσά και νούμερα. Γιατί εμεί είμαστε Επιτροπή Προπολογισμών. Χωρί αριθμητικά ποσά δυσκολευόμαστε να λειτουργήσουμε. Παρακαλώ να το έχετε υπόψη αυτό και να το εξασφαλίζετε στο μέλλον. Δεύτερον, έχω μια παράκληση για το κτίριο Τάντενα, ο ΕΡΚΑΤ, στο Λουξεμβούργο. Ε, θέλω να έχουμε μια καλύτερη εικόνα και πιο ακριβή. Τι έγινε τώρα, τελείωσε το εργοτάξιο, πόσο κόστισε, πόσο κόστισε κάθε τι, για να έχω και τη δυνατότητα να μελετήσω τι αποφάσισε η Επιτροπή Προπολογισμών, τι προσθέθηκε επιπλέον για λόγους ασφαλείας κλπ. Και τι γίνεται με την ε, τελευταία ε, ε, εικόνα, την κατάσταση πραγματικά. Ε, θέλω να ευχαριστήσω πολύ και να συγχαρώ τον κύριο Βίλαντ για τα νέα γραφεία. Είδα τις νέες δυνατότητες που έχουμε και σε σχέση με αυτό που έχουμε μέχρι τώρα είναι κβαντικό άλμα αυτό, όχι ποιοτικό. Και ε, επίσης είναι πολύ θετικό αυτό. Μιλήσαμε για την ε, ε, κουλτούρα επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων στα νέα κτίρια, ακριβώ το ίδιο χρειάζονται και βουλευτέ. Δηλαδή χρειάζεται να έχουμε χώρου. Ε, στο 13ο και στο 14ο όροφο όπου έχουμε ένα γραφείο γυάλινο που μπορεί κανείς να πάει ε, εύκολα και γρήγορα για να κάνει και μια σύσκεψη ας πούμε όταν θέλεις να έχεις μια συνεργασία με 7 συναδέλφους, πηγαίνεις γρήγορα σε ένα τέτοιο γραφείο και κάνεις ε, μια συνάντηση με ειδικού εμπειρογνώμονες και δεν ε, χρειάζεται ε, να γίνεται αυτό σε κατάσταση πολιορκίας σε διάφορα γραφεία. Είναι θετικό αυτό και το ύφο είναι θετικό και το στυλ των επίπλων, γιατί δεν είναι από τη δεκαετία του 70, ας πούμε, σαν αυτά που έχουμε τώρα. Και δεν είναι όλα τετράγωνα, ξέρω εγώ, γυάλινα, σιδερένια, ε, ε, που είναι ε, παλιά στα γραφεία μας και χρειάζεται και λίγο να τα συνηθίσει κανείς. Ξέρετε την παλιά διαφήμιση για μια γερμανική σοκολάτα που ήταν το σλόγγαν τετράγωνο πρακτικό καλό. Δεν είναι πάντα αυτό καλό το τετράγωνο και το πρακτικό. Λοιπόν, έχουμε νέες δυνατότητες ε, για καλύτερη επικοινωνία, ταχύτερη επικοινωνία και ε, ευκολότερη. Το θέμα της συστηματικής πολιτικής ανακαίνησης των κτηρίων θεωρώ άκρο σημαντικό. Ε, το βλέπουμε αυτό στους δύο πύργους με τα γραφεία των βουλευτών. Ξέρετε κάθε πόσο χαλάει το καρυματιστικό. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τη συντήρηση και όταν χτίστηκαν τα κτίρια δεν ήταν η σημερινή προδιαγραφή. Στο δικό μας 15ο όροφο, για να το πω έτσι κομψά, κάθε μέρα παραμέρα ένα χοντρό καλώδιο κάποιου σερβερ ε, μας ρίχνει το κλιματιστικό. Ε, οπότε εκεί χρειάζονται και μέτρα συντήρησης και μέτρα ανακαίνησης με το σωστό και κατάλληλο τρόπο. Επίσης έχουμε και το πρόβλημα με τη λεγιονέλα και τα λιμνάζοντα ύδατα ε, και βλέπουμε κάτι περίεργα πλαστικά ντους του παρελθόντος που υπάρχουν ακόμα. Είναι προβληματικό αυτό και για την υγεία και για την ε, ασφάλεια των ανθρώπων και την πρόνοια για αυτούς που εργάζονται σε αυτά τα γραφεία. Στρασβούργο και Βρυξέλλες. Χαίρομαι πολύ που θέλετε να μας δώσετε ένα συνένα γραφείο. Το Χάβελ αποφασίστηκε στην περασμένη θητεία και τώρα ε, διαμορφώνεται κατάλληλα και το λέω προς την κατεύθυνση όλων που, εκείνων που επιθυμούν ε, τη μία ενιαία έδρα, ότι ωραίο είναι αυτό που το ψηφίζουμε εμείς, αλλά μας αγνοεί το Συμβούλιο και θα ξεκολουθήσει να μας αγνοεί για την επόμενη δεκαετία, οπότε πρέπει να κάνουμε και τη δουλειά μας. Για το κτίριο PHS Polaris Park έχω μια συγκεκριμένη παράκληση. Πριν αρχίσουμε να το συζητάμε με πολίτες διάφορους, καλό θα ήταν να μας ενημερώσετε για να μην τα μαθαίνουμε από τον τύπο. Είναι τα μέσα ενημέρωσης από την πρωτοβουλία πολιτών. Γιατί από αυτή τροφοδοτούνται ε, τα μέσα ενημέρωσης και είναι απόψεις διαφόρων έτσι, προσωπικές. Αφού ε, είχα την ευκαιρία να κοιτάξω έγγραφα για το κτίριο PHS, ε, οφείλω να πω ότι μου κάνει εντύπωση και μόνο που πήρε την άδεια να χτιστεί ένα τέτοιο κτίριο εκεί που βρίσκεται, αλλά τώρα το έχουμε και να κάνετε πραγματικά ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι πρέπει να γίνει και πότε. Έχω και μια ερώτηση για το λεγόμενο κτίριο Belmont. για το Μοντουαγέ 63 προσωρινά έχει αντικατασταθεί από το κτίριο Belmont. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο αριθμητικό και οικονομικό ε, στο έγγραφο εργασία και πάλι δεν αναγράφονται πουθενά ποσά. Γράψτε και κανένα νούμερο κάποια στιγμή, γιατί γι' αυτό έχουμε τα έγγραφα εργασία για να κάνουμε τη δουλειά μα. Μετά υπάρχει επιλογή αγοράς για το ΤΡΕΒ και το μοντοαγέ 75. Παρακαλώ να μας ενημερώσετε για το πώς βαίνουν οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή των συμβάσεων. Σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Βίλαντ για το κτίριο στο Παρίσι, και όλα τα γραφεία ενημέρωσης. Έχω και εγώ την ίδια εντύπωση με τον κύριο Βίλαντ και δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω και να τονίσω αυτό που είπε και ο ίδιος. Το συζήτησα και με τον αρμόδιο επίτροπο για τον προϋπολογισμό και παρακαλώ να έχουμε μια γενική κατανομή και να μην μετράμε κάθε τετραγωνικό, αλλά μισά-μισά όλα τα γραφεία. Και να συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οικονομικά ε, στα κτίρια που χρησιμεύουν για την προβολή και παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην τσακωνόμαστε κάθε φορά για τα κτίρια. Και ή δυνατόν τα κτίρια να μην είναι στην τελευταία ανθυποπάροδο που δεν περνάει ψυχή απ' έξω, αλλά σε χώρους με μεγάλη κυκλοφορία και με αυτόματη προσέλευση του κόσμου. Τα άλλα κτίρια δεν ήταν κακά τα ίδια, αλλά ήταν στο πουθενά. κόσμος δεν αντιλαμβανόταν τι υπάρχει εκεί και για να πάει κάποιος επισκέπτης έπρεπε να πάει ειδικά, δηλαδή να ενδιαφέρεται οπωσδήποτε για το γραφείο του Κοινοβουλίου, να το ψάξει, να το βρει, ε, πού βρίσκεται στο χάρτη και να πάει να μπει μέσα. Και οι νέες λύσεις, ε, είτε πρόκειται για το Βερολίνο, το Παρίσι και τα λοιπά, είναι πολύ καλύτερες. Γιατί είναι αυτόματα ε, σε χώρους που κυκλοφορούν τουρίστες ή και ντόπιοι και είναι εξέχουσα θέση και προβεβλημένη και μπαίνει ο κόσμος. Αυτά προς το παρόν, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Συγγετρία. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα τους και οδησηγητές, τους παρόντες αν με τι άλλο. Ο κύριος Ντιπχέ είναι ο πρώτος, Ζεγάχ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη γιατί υπάρχουν προβλήματα κυκλοφορίας και έφτασα με καθυστέρηση και δεν άκουσα το σύνολο των προηγούμενων παρεμβάσεων. Τρία σχόλια. Χαίρομαι για αυτήν εδώ τη συνάντηση. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε για τα κτίρια. Μια παρατήρηση επισκέφθηκα με αρκετή καθυστέρηση το νέο κτίριο Μάρτενς. Νομίζω ότι πράγματι πρόκειται για ένα ωραίο κτίριο, έχει σχεδιαστεί σωστά και νιώθει κανείς ε, ωραία. Να πω κάτι το χιδαίο λίγο. Ε, δεν υπάρχουν ε, βέβαια τέτοιου είδους κτίρια με αυτό το επίπεδο ποιότητας, συνεπώς την καλοπιάνεται τη διοίκηση του Κοινοβουλίου και τους υπαλλήλους ε, να σας βάλω να επισκεφθείτε τα γραφεία μου στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες για να καταλάβετε τη διαφορά αντιμετώπισης που υπάρχει ανάμεσα στους βουλευτές και τους υπαλλήλους. Φυσικά οι βουλευτές είναι περαστικοί, αλλά αυτός δεν είναι λόγος έτσι ώστε συστηματικά να μας περιφρονείτε. Εξετίμησα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σασόλη σχετικά με τον σεβασμό των ενεργειακών κανόνων. Αν κατάλαβα επίσης καλά, αυτά τα οποία είπια, είπαν κάτι, δεν ξέρω ποιος το είπε, αν το είπε ο κύριος ε, Βέλε ή ο κύριος ε, Βίλαντ, το Προεδρείο φαίνεται ότι θέλει να δημιουργήσει ένα παρλαμαντάριο σε κάθε κράτος μέλος. Κατάλαβα καλά. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Σε όλα τα κράτη-μέλη δηλαδή τώρα από εδώ και πέρα θα έχουμε ένα γραφείο του Κοινοβουλίου, μια επίσημη υπηρεσία του Κοινοβουλίου και ένα παρλαμεντάριο. Τώρα μήπως θα μπορούσαμε να εναρμονίσουμε τα δύο έτσι ώστε να μην υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους επενδύσεις σε κάθε μία από τις χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ακριβώς έχετε σκεφτεί γύρω από αυτό το, αυτή τη στρατηγική επιλογή. Ήσασταν πάρα πολύ σύντομοι και ίσως έλειπα και πιο πριν εγώ. Το θέμα είναι το πιο ευαίσθητο και ομιλώ ως Βέλγος. Και ξέρω ότι πολλές φορές ε, λέγεται ότι στο Βέλγιο δημιουργούν κτίρια τέρατα και θα απαντούσα σε αυτούς ότι αν η μια γειτονική μας χώρα ήταν τόσο θαυμάσια αρχιτεκτονικά κάθε Σαββατοκύριακο θα πηγαίναμε να το δούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει για το PHS, ε, το τι θα κάνουμε με το PHS αν τυχόν πάρουμε την απόφαση να χτίσουμε ένα νέο κτίριο είναι μία απόφαση που και οικονομικά και πολιτικά θα έχει τρομακτικές συνέπειες. Οι πολίτες βλέπουν το τι γίνεται σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι πολίτες πιστεύουν ότι οι ευρωβουλευτές ζουν πολύ καλά, καμία σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες και αν τυχόν χτίσουμε ένα νέο κτίριο, η επιχειρηματολογία μας θα πρέπει να είναι θωρακισμένη θα έλεγα. όχι μόνο το κτίριο λοιπόν να είναι θωρακισμένο, αλλά και η επιχειρηματολογία. Κατανοώ λοιπόν αυτά τα οποία υπόθηκαν, αλλά οι επιλογές είναι δύο πλέον. Ή μία μίζων αναδιαρρύθμιση ή ε, ένα νέο κτίριο με προκήρυξη για τη σχεδίαση κτλ. Αν το αποφασίσουμε αυτό πριν από τις επόμενες εκλογές, θα πρέπει τα επιχειρήματα να είναι ισχυρά. Γιατί τη στιγμή κατά την οποία ένας μεγάλος αριθμός των πολιτών διαρωτώνται για το αν θα πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε την Ευρώπη, εμείς δώσουμε την εικόνα ανθρώπων οι οποίοι ε, δεν ενδιαφέρονται παρά για τη φιγούρα θα έλεγα και τους μισθούς τους. Ε, εγώ είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι το θέμα αυτό θα μπορούσε να έχει αποσταθεροποιητικές συνέπειες σε ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος. Πριν ληφθεί λοιπόν απόφαση για διαγωνισμό θα πρέπει όλοι οι ευρωβουλευτές και ιδιαίτερα εμείς εδώ να έχουμε επιχειρήματα στη διάθεσή μας που θα μας επιτρέψουν να προασπιστούμε την επιλογή αυτή. Guardia που αντικαθιστά τους και ηγητέ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τους αντιπροέδρους και το Γενικό Γραμματέα που ήρθατε να μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες. Όλοι γνωρίζουμε ότι η διαχείριση ε, της κτηριακής πολιτικής είναι και περίπλοκη, αλλά και τα τελευταία χρόνια, μάλλον πριν από 15 και 20 χρόνια δεν ξέραμε τι ανάγκες είχαμε. Τώρα που ξέρουμε, δεν είναι καθόλου προφανές τι πρέπει να κάνουμε, αλλά στις αποφάσεις που θα πάρουμε από εδώ και στο εξή θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τρεις μεταβλητές, ας πούμε, τις ανάγκες, το κόστος και τη χρήση και τη χρησιμότητα. Εγώ κάνω μεγάλη ε, διαφορά στι δύο προτάσει για τα κτίρια στι Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Είναι προφανή οι ανάγκε ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χώρο για να δουλεύουμε πιο άνετα και εμεί και οι συνεργάτε μα. Αλλά στι Βρυξέλλες ε, χρησιμεύουν πολύ περισσότερο τα γραφεία από ό,τι στο Στρασβούργο. Και μιλάω από την προσωπική μου πείρα φυσικά στο Στρασβούργο. Περνάμε στο γραφείο μία ώρα τη μέρα, γιατί όλη μέρα έχουμε συνεδριάσεις. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε στο Στρασβούργο είναι ότι δεν έχουμε στη διάθεσή μας μικρές αίθουσες για να ε, συνεδριάζουμε τον κόσμο που υποδεχόμαστε στο Στρασβούργο. Ε, και θα έβρισκα πολύ πιο οικονομικό, πολύ πιο αποτελεσματικό και πιο χρηστικό, βάση περιπτώσει, να ε, ψάχναμε αίθουσε πολλαπλών χρήσεων που να μπορεί κάποιο να κλείνει online, να κάνει τη δουλειά του αντί να διπλασιάσουμε το χώρο των γραφείων. Άλλες ανάγκε έχουμε στις Βρυξέλλε και άλλες στο Στρασβούργο. Και κυρίως, γιατί εντό εισαγωγικών αυτό είναι και ίσον σημασία θέμα, να μην ξαναβρούμε μπροστά μα αυτό που είδαμε στο CAD, να έχουμε ένα CAD 2. Εγώ είμαι εδώ δυο θητείες και είναι το γεφύρι της άρτας. Δεν ξέρω ούτε πόσα χρήματα έχουμε ε, δαπανίσει, πόσες φορές έχουμε αλλάξει το σχεδιασμό και πότε θα τελειώσει και πόσο θα κοστίσει. Για το Polaris Pack. Άκουσα από τον κύριο Τεμπρέ κάτι διαφορετικό. Μάλλον κατάλαβα εγώ κάτι διαφορετικό από τον κύριο Τεμπρέ. Ότι έχουμε δύο επιλογές και θα κάνουμε ένα διαγωνισμό για να δούμε ποια έργα είναι βιώσιμα και τι κόστος ε. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση η εκτίμηση των δύο επιλογών. Ότι είναι τόσο ακριβή η ανακαίνιση σε σύγκριση με την κατεδάφιση και ανέγερση νέου κτηρίου. πολύ μεγάλη η διαφορά. Φυσικά δεν είμαι ειδική, αλλά και κατανοώ ότι είναι πολύ ακριβό να ανακαινήσεις ένα κτίριο. Αλλά να κοστίζει περίπου το ίδιο με το να το γκρεμίσει και να χτίσει ένα καινούριο, με εκπλήσει αν μη τι άλλο. Δεν ξέρω αν έχετε επιπλέον πληροφόρηση. Ευχαρίστω. Και συμφωνώ με τον κύριο Ντεπχέ. Η απάντηση για το ε, PSS ε, είναι πολύ σημαντική οικονομικά και πολύ λεπτή και ευαίσθητη πολιτικά. Θα, πρέπει να έχουμε πολλές προφορίες, ε, όλα τα στοιχεία και να πάρουμε την ε, απόφαση με ηρεμία. Αυτό για το 3% υπάρχει ε, ένας προγραμματισμός ή τώρα το προγραμματίζεται. Ε, όχι μόνο τη δράση αλλά και τη χρηματοδότηση. Να ξέρουν αυτοί που θα είναι εδώ τα επόμενα χρόνια σε ποιες δαπάνες μπαίνει το, ο προεπιλογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ως γενική παρατήρηση θα πρέπει τέτοιου είδους ανταλλαγή απόψε να έχουμε πιο συχνά γιατί καλούμαστε να αποφασίσουμε για ε, τον προϋπολογισμό και πολλές φορές μας έρχονται από το Προεδρείο έτοιμες οι ε, αποφάσεις και εμείς θα πρέπει να βάλουμε μόνο μια σφραγίδα προς πληρωμή. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα τέτοιες συνεδριάσεις για ενημέρωση, για συζήτηση και τροποποίηση ενδεχομένως κάποιων προτάσεων που συζητάει το Προεδρείο. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Vous en prie. Okay, I'm sorry. Λοιπόν, κατανοώ ότι στις σημερινές συζητήσεις ο Γενικός Γραμματέας ε, Βέλε θα θυμάται για πάντα κάθε πρωί που ε, στεκόταν μπροστά στον καθένα και έπρεπε να έρθει στην Επιτροπή προπολογισμό και να μας ε, μιλήσει. Υπήρξαν όμως κάποια ερωτηματικά όσον αφορά το σχέδιο να γκρεμίσουμε το PHS γιατί αναφέρεται ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι 25 έτη και αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να εξηγήσω ακόμα και στον εαυτό μου ότι χτίζουμε με ένα τέτοιο τρόπο ακόμα και μια αναπηρική καρέκλα αναπηρικό μαξίδι κρατάει περισσότερο καιρό. Είναι δύσκολο λοιπόν να το εξηγήσουμε και γι' αυτό προτείνω να αναβάλουμε τα σχέδια για μετά τον Μάιο του 2019. Δεν είμαι εδώ. Δεν είμαι εδώ τότε για να εξηγήσω αυτέ τι πολιτικέ, τι κτηριακές Και ένα σημείο στο οποίο διαφωνώ με τον κύριο Ντεπάε, που είπε ότι τα μέλη ε, ότι δεν ε, έχουν ε, σωστή μεταχείριση όσον αφορά τις εργασιακέ συνθήκες τα πιο πολλά πιο πολλοί ευρωβουλευτές είναι από την Ανατολική Ευρώπη. Και εδώ η κατάσταση έχει βελτιωθεί αρκετά. Ενδεχομένως να μην υπάρχουν ε, επαρκή τετραγωνικά μέτρα και τα λοιπά για τους βοηθούς και όλα αυτά. Αλλά ίσως θα έπρεπε να αναγνωρίσουμε ότι και οι βουλευτές και οι βοηθητούς δεν είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν τα, τις χειρότερες συνθήκες στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γκαγιέρ. Γκάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω όσον αφορά τη ρυθμίση των γραφείων. Είμαι, το γραφείο γνώμων. Θα μου άρεσε αν θα πιο μοντέρνη ιστορική αρχιτεκτονική. Με το μέγεθο κάτι κάναμε. Όταν ήρθα το 2009 μου έκανε εντύπωση ότι, ότι βρήκα ένα υγρό δωμάτιο Το ντους δεν λειτουργούσε στο διαμέρισμά μου Άρα είναι κάτι που χρησιμοποιείται από τους ε, βουλευτές, τον ντουζ αυτό. Ε, επίσης έκανα μπάνιο στο γυμναστήριο. Υπήρχε μια ξαπλώστρα ουσιαστικά όπου μπορούσε κανείς να ξαπλώσει, μετά έγινε καναπές. Όσον αφορά το PHS, ένα πράγμα με προβληματίζει. Δεν συμφωνώ με τον ξέρουμε, συνάδελφο Βίλεν. Κάθε 30 χρόνια θεωρώ ότι ένα τέτοιο κτίριο χρειάζεται μια ενεργειακή αναβάθμιση και ότι θα πρέπει να ανακαινιστεί. Το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό που δεν μπορώ να εξηγήσω εύκολα είναι το ότι πρέπει να γκρεμιστεί τέτοιο κτίριο, όπως πήγε ο συνάδελφος. Καταλαβαίνω λίγα από αυτή δηλαδή αλλά πολλά από επικοινωνία. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα με τέτοιου είδους εικόνες. την ε, ε, διάδοση της ιδέας της ολοκλήρωσης της Ευρώπης. Θα πρέπει όλα να είναι αποδοτικά προς το κόστος, αλλά να μην έχουμε και... Ε, να μην έχουμε μια κάποιο είδους δυσήμιση σε περίπτωση θα γκρεμίσουμε το κτίριο PHS. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στους τρεις προσκεκλημένους μας, θα ήθελα να επιμείνω επί ενός σημείου που έθεσε η Μόνικα Χόλμο για την ενημέρωση δηλαδή σε επίπεδο δημοσιονομικό. Με τον Τιν Λαού οργάνωσα μία συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα γιατί στο όνομα της εμπιστευτικότητας για τα θέματα της ασφάλειας σας ζούμε σε μία απουσία ενημέρωσης. Η κατάσταση αυτή δεν θα συνεχιστεί. Εμείς πρέπει να έχουμε οικονομικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να επανέλθω σε σχέση με την τήρηση ή μη αυτής της αρχής. Αναφερθήκατε επίσης στο PHS και για το αν θα πρέπει να, να, ε, να χτίσουμε ένα καινούριο κτίριο. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της περίοδου εν πάση περιπτώσει ε, που θα κρατήσει ε, η διαδικασία το Στρασβούργο θα ήταν μια καλή λύση. Και πέραν αυτού, κύριοι Πρόεδροι και κύριε Γενικέ Γραμματέα, μπορείτε να μας δώσετε κάποια επιπλέον στοιχεία απάντησης. Ο κύριος Βίλαντ, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θέλω κάτι να συμπληρώσω. Μην τυχόν και βγει κανένας ε, διαμαρτυρόμενος ότι εκπλήσεται. Ότι δεν έχουμε ανάγκες στο Στρασβούργο. Μα εμείς είμαστε στραμμένοι προς το μέλλον. Ε, για τα θέματα ασφαλείας, α πούμε, στο Στασβούργο χρειάζεται δουλειά. Λοιπόν, μην εκπλακείτε ε, που θα δείτε κάποια πράγματα. Κύριε Ντεπρέ, ε, όταν ήρθατε είχα μιλήσει και πριν έρθετε πραγματικά μπορώ να σα διαβεβαίωσω είπα κάποια πράγματα με τα οποία θα είστε απολύτως σύμφωνο, και μην ανησυχείτε. Να σας πω δύο περιστατικά. Πρώτον, πριν από δύο χρόνια υπήρχε μια σκέψη, δυόμιση τώρα δεν θυμάμαι, τι θα κάνουμε, ε, τι κάνουμε με, τα έπιπλα, με τον εξοπλισμό μας μετά από 25 χρόνια. Οι περισσότεροι είπαν ότι ανακλαστικά δεν τα χρειαζόμαστε. Ε, δεν τα προσέχουν όλοι ε, όσο οι περισσότεροι από εμά και χαλάνε. Και τώρα βλέπουμε τι δυνατότητα υπάρχει και όλοι λένε καλή λύση αυτή. Να μην τα επισκευάσουμε, να τα αλλάξουμε. Δεύτερο περιστατικό, το κτίριο Μάρτενς. Θυμάστε την ιστορία με το New York ε, World of ε, World of Work ε, οι πολλοί είχαν ε, μεγάλες επιφυλάξεις και τώρα έχουμε στο Μάρτενς ε, μια εφαρμογή light και είμαι ικανοποιημένο και το έχουν δεχτεί και οι υπάλληλοι. Αλλά πριν από τρία χρόνια ε, υποδίονταν οι ότι, ότι θα χρειαστούν να τους μαστιγώνουν για να μπουν στο κτίριο και τώρα κάνουν ουρά. Εκείνοι που κατήγγυλαν παγκόσμιες συνωμοσίε. τώρα ε, είναι πάρα πολύ ταπεινοί μπροστά στη νέα κατάσταση. Η κυρία Γκόρδια Σαμπάλ μίλησε για το κτίριο ΚΑΔ στο Λουξεμβούργο. Εγώ είμαι στο πρόεδρο από το 2009 και ήρθα μπροστά σε τετελεσμένα κατά κάποιο τρόπο. Και μου είπαν πώς πήγαν τα πράγματα, ότι ήταν πάρα πολύ φιλόδοξος ένας πράσινος αντιπρόεδρος και είχε προτείνει στο Κοινοβούλιο κάποια πράγματα που θα είχαν κάποια περιβαλλοντική τεχνολογία ε, στο μέλλον, τα οποία όμως ποτέ δεν υλοποιήθηκαν γιατί δεν έφτασαν στην αγορά αυτές οι προτάσεις τεχνολογικές. Και μετά, ε, επειδή φοβόντουσαν τα μεγάλα ποσά, άρχισαν να χτίζουν πριν ολοκληρωθούν τα σχέδια. Μα τι θέλουμε τώρα. Δεν μπορούμε να έχουμε για 4, 6, 8 σενάρια ε, τιμολόγηση μέχρι τελευταίο ευρώ μας κοστίζει και αυτό μεγάλα ποσά. Γιατί θα έχουμε 4, 6, 8 διαδικασίες παράλληλα. Τώρα το Κοινοβούλιο λέει να το περιορίσουμε σε δύο επιλογές. Με ανοιχτή έκβαση. Και ήρθανε παράπονα ε, ε, και καταγγελίες, κύριε Γκάιερ. Δεν θα ήταν καλή δουλειά κάποια πράγματα τα λέγαμε δημόσια. Γι' αυτό σας δεν παραπέμπω στον αγνωστήριο. Και περιμένω ε, κάθε πολιτική ομάδα να έχει στείλει ένα μέλος της στον αγνωστήριο. Γιατί, κυρία Κορδιά Σάμπα, γιατί είναι τόσο ακριβή σχετικά η ανακαίνιση σε σύγκριση με την ανοίγερση νέου κτηρίου. Τα λέει ο πυρογνώμονας αυτά. Λέει ότι κοστίζει απίστευτα ποσά στην ανακαίνιση να καλύψουμε τα ελλείμματα που έχει στην ασφάλεια το κτίριο και είναι σαφή. Με την ανακαίνιση είναι αρκετά τα χρήματα και δεν μπορεί και να μας εγγυηθεί κιόλα ότι θα είναι σε επίπεδο ασφαλείας το κτίριο το οποίο σήμερα θα συνιστούσε. Γι' αυτό αν πάτε στο αναγνωστήριο θα το καταλάβετε. Αλλά μέσα είμαστε κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε να δώσουμε λαβή έτσι ώστε διάφοροι στο διαδίκτυο να κυκλοφορούν οδηγίες χρήσεως και κατασκευής διαφόρων πραγμάτων. Γι' αυτό σας λέω, όχι δημόσια, αλλά ε, να τα διαβάσετε. Και για την πρωτοβουλία πολιτών που ακούστηκε. Το διάβασα κι εγώ αυτό το άρθρο. Φοβερό άρθρο, το οποίο αναμειγνύει με τρόπο δόλιο θα έλεγα. Και έτσι υποχθώνει ότι γίνεται με το κτίριο Βίρτς, ε, το σπίτι δηλαδή του καλλιτέχνη ε, και το αναμειγνύει πάρα πολύ ε, ωραία και έντεχνα με τις εργασίες που γίνονται στο κτίριο Πολαρή Σπακ. Για το, την αίθουσα αυτή, τη γυάλινη, πραγματικά κάποια στιγμή την ανακάλυψα και χρειαζόμαστε Μάλλον έχουμε 15 τέτοιους χώρους που δεν τους χρησιμοποιούμε. Είναι κάποιες γυάλινες αίθουσες. Και τι θέλω στο μέλλον, εσωτερικές δηλαδή, να έχουμε καλύτερο σύστημα κράτησης αιθουσών. Ε, οι πολιτικές ομάδες, ο πρόεδρος και άλλοι έχουν δυνατότητες. Αν ο καθένας κάνει λίγο πίσω ε, θα έχουμε συνέργειες. Αλλιώς, αν περιχαρακωθεί ο καθένας στα τετραγωνικά που έχει και δεν κάνει σπιθαμή πίσω, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η σύγχρονη κτηριακή πολιτική, να έχουμε μικρές αίθουσε ευέλικτα, να μπορούμε να τις ε, κρατάμε online και να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα με μεγαλύτερη οικονομία. Ευχαριστώ κύριο Σασόλη. Σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε να σας ευχαριστήσω όλους για τις παρατηρήσεις τις οποίες κάνατε και σχετικά με αυτά που είπα και σχετικά με αυτά που είπαν ε, ο συνάδελφος Βίλαν και ο γραμματέας Βέλε. Κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη για διάλογο εμείς είμαστε διαθέσιμοι και αυτό εξαρτάται κυρίως από εσά, από τη δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Σε ό,τι μας αφορά όμως δεν έχει υπάρξει κανένα πρόβλημα. Για τον χρονισμό. Αν εμείς οικοδομήσουμε ένα νέο κτίριο, δεν θα το κάνουμε αυτό όπως το είχαμε κάνει 20, 30 ή 40 χρόνια στο παρελθόν. Το Μάρτενς είναι ένα παράδειγμα. Το Μάρτενς δεν είναι μόνο θέμα διαρρύθμισης, αν έχετε μια κάποια περιέργεια πηγαίνετε να δείτε τι υπάρχει πίσω από το Μάρτενς. Δηλαδή στις αίθουσε των μηχανισμών που τον μηχανολογικό εξοπλισμό για το ζεστό νερό, τη θέρμανση, την ψήξη. Το σύστημα είναι πρωτοπόρο και είναι ένα σύστημα το οποίο διαπνέεται από μια καινοτόμο λογική εξοικονόμησης ενέργειας. Είναι προφανές ότι αυτό το οποίο φτιάχνουμε σήμερα δεν το κάνουμε λοιπόν όπως πριν 20-30 χρόνια. Για το PHS. Πολλοί είπανε γι' αυτό. Το PHS έχει σημαντικά προβλήματα. Να σας πω κάποια από αυτά ηλεκτρική εγκατάσταση, υδραυλική εγκατάσταση, παλαιότητα κάποιων υποδομών, κατανομή των χώρων, η οποία δεν επιτρέπει να έχουμε την επιθυμητή λειτουργικότητα, αίθουσες για τριγωνικούς διαλόγους κτλ μια χωρική διανομή που δεν μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλους τους χώρους όπως θα θέλαμε. Είχαμε επίσης και το θέμα της ασθένειας των... για την ασθένεια των λεγεωναρίων με τα στάσιμα θερμαίδατα σταθερότητα της ε, οροφής της Ολομέλειας. Έχουν γίνει πολλές τεχνικές παρεμβάσεις ε, στο άνω μέρος. Είχαμε επίσης προβλήματα αιθουσών γιατί δεν υπάρχουν πολλές αίθουσες μικρών διαστάσεων και κάθε φορά που κάποιος χρειάζεται μία αίθουσα παίρνει μία αίθουσα 20-30 ατόμων. Είχαμε προβλήματα επάνδρωσης ε, αν θέλετε των αιθουσών, εξοπλισμού των αιθουσών για την διερμηνία ε, και το PHS παρουσιάζει λοιπόν πάρα πολλά προβλήματα. quattro le Quella di non fare... Έχουμε λοιπόν δύο δυνατότητες. Ή να μην κάνουμε τίποτα ή να προχωρήσουμε στην αναδιαρρύθμιση του κτηρίου ή να προχωρήσουμε στην επανικοδόμηση, λέει ο μιλητής και επίσης θα μπορούσαμε να κάνουμε μια επιμέρους αν θέλετε ανακαίνιση. Εμείς λοιπόν τι αποφασίσαμε. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί. Ας μειώσουμε τις επιλογές και ας προσπαθήσουμε να τις κατανοήσουμε καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάναμε μία επιλογή. Εγώ προσωπικά, όπως και πολλοί από εσά, πρέπει κάνουμε ότι πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι γίνεται για να ανακαινήσουμε. Και για λόγους εικόνας του Κοινοβουλίου, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, το πρόβλημα της επικοινωνίας αυτής της παρέμβασης είναι πάρα πολύ ευαίσθητο σε σχέση με την κοινή γνώμη. Εάν όμως πράγματι θέλουμε να πάρουμε μια σοφή απόφαση, θα πρέπει να κάνουμε πρώτα κάποιες εκτιμήσεις, αξιολογήσεις. Αποφασίσαμε λοιπόν να μειώσουμε σε δύο τις επιλογές και να εμβαθύνουμε στις επιλογές αυτές δεν θα πάρουμε την απόφαση αυτή κατά τη διάρκεια της ε, παρούσης κοινοβουλευτικής ε, περίοδου. Θα χρειαστεί χρόνος και για τις μελέτες πιο αναλυτικά. Ο καθένας θα μπορούσε να είναι υπέρμαχος ιασδήποτε επιλογής. Αλλά τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε αν δεν λάβουμε υπόψη μας τεχνικά, αντικειμενικά και επαγγελματικά ελέγξιμα και κατάλληλα στοιχεία και τότε μόνο μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις. Γι' αυτό λοιπόν και αποφασίσαμε υπεύθυνα να κάνουμε την πρόταση αυτή και να καταστήσουμε τους πάντες ικανούς να συμμετέχουν σε μια δημόσια συζήτηση αλλά με αντικειμενικά κριτήρια. Ευχαριστώ κύριε Σασόλη, κύριε Γενική Γραμματέα πάρα πολύ σύντομα διότι έχουμε καθυστερήσει ιδιαίτερος. Η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα άλλωστε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα περιοριστώ στην προσπάθεια να απαντήσω ερωτήσεις και χωρίς να σχολιάσω. Ε, ε πρώτη ερώτηση κυρία Σχόλμαγερ για το κόστος του κτηρίου Belmont. 1,44 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ακριβώς το ίδιο ποσό που ε, καταβάλαμε για το κτίριο μέχρι τώρα, το άλλο, το Μοντουαγέ με το ίδιο ποσό μας δίνουν αυτό το κτίριο προσωρινά προς αντικατάσταση. Ο κύριος ε, Ντεπρέ είπε ότι το κτίριο Μάρτες είναι καλύτερο ε, για τη διοίκηση από ότι για τα κτίρια για τους βουλευτές. Έχουμε διαφορά στην αρχιτεκτονική 30-40 ετών και στην τεχνολογία για το πώς μπορεί κανείς να επικοινωνεί. Το κτίριο Μάρτενς είναι το πρώτο κτίριο που έχουμε όπου έχουμε σκεφτεί συστηματικά πώς θα επικοινωνεί ο κόσμος καλύτερα. Μέχρι τώρα στα γραφεία των βουλευτών αυτό τελείως ε, ε, ανεπαρκώς έχει γίνει και μέσω πρόθεσμα θα πρέπει αυτό να έχει επιπτώσεις και για τους χώρους των βουλευτών. Ο Αντιπρόεδρος Βίλαντ ε, ε, για κάποιες αίθουσες και κάποιους χώρους. Προς τα εκεί κινούμαστε. Ο κύριος Ντεπρέ επίσης ρώτησε κάτι για το θέμα Experience Europe. Ε, ναι, το Προεδρείο αποφάσισε σταδιακά την επόμενη δεκαετία ε, αυτό να γίνει και στα εξωτερικά γραφεία, ένα είδος παρλαμεντάριο. είναι ένας τομέας μόνο Ας πούμε στη Σλοβενία υπάρχει αυτό, είναι πάρα πολύ μικρός χώρος στη Λουμπλιάνα, αλλά μπορεί να έχει και μεγαλύτερες διαστάσεις και έκταση ανάλογα με τη χώρα και τους χώρους που έχουμε εκεί. Η κυρία Γουαρδιά ρώτησε ε, τι γίνεται με το κόστος του PHS βασικός ε, στόχος αυτού του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού είναι να έχουμε πιο αξιόπιστους υπολογισμούς για το κόστο. Μέχρι τώρα είναι πολύ αφηρημένα όλα αυτά. Με το συγκεκριμένο διαγωνισμό ε, ελπίζουμε να μας κοστολογήσουν αυτές τις δύο δυνατότητες ε, με ακρίβεια και τι θα αποκομίσουμε από την κάθε επιλογή για να αποφασίσει το Προεδρείο Μεταλόγου Γνώσεως και η Επιτροπή Προεπολογισμών για τα ποσά. Κύριος Τάραντ αναφέρθηκε και πάλι στο κτίριο PHS. Κοιτάξτε, δεν το χτίσαμε εμείς. Το κληρονομήσαμε, δηλαδή το, το αγοράσαμε εκ των υστέρων, ήταν ήδη εκτισμένο. Ο κύριος Γκάιε είπε ότι χρειαζόμαστε νέο εξοπλισμό οπωσδήποτε για τους βουλευτές ε, έπιπλα δηλαδή. Και μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα σε λογικές τιμές. Ευχαριστώ για τη συντομία σας κύριε Γενικέ. Ε, κύριε Ντεπρέ, συμπροματική ερώτηση. Συζητώ συγγνώμη κύριε Βέλε. Έκανα μια συγκεκριμένη ερώτηση. Το Προεδρείο έλαβε νέου απόφαση να ε, ε, φτιάξουμε παρλαμεντάριο σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης και προβλέπεται αυτό το παρλαμεντάριο να συνδέεται με τα γραφεία του συνδέσμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διάφορες χώρες. Απάντησε. Θα απαντήσω γαλλικά. Δεν θέλω να κατηγορήσω τους διερμηνείς, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω στα γαλλικά. Μάλιστα, αποφάσισε το Προεδρείο να σκεφτεί να δημιουργήσει αυτή την εμπειρία Ευρώπη που είναι κάτι διαφορετικό από το Παρλαμεντάριο σε όλες τις χώρες. Αυτό το Experience Europe αλλά μόνο αφήστε, όταν έρθει η ώρα να θεώρησε το συμβάσεων. Δεν γίνεται αυτό αυτόματα του χρόνου σε δύο χρόνια, αλλά σταδιακά ε, και από αυτό μπορεί να πάρει μια δεκαετία και παραπάνω. Δεύτερον, Αυτές οι εγκαταστάσεις λοιπόν θα είναι στα γραφεία ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θα έχουμε διαφορετικούς χώρους, θα είναι ε, ε, ε, μία από τις δραστηριότητες του γραφείου αυτού για την ενημέρωση του κοινού. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ και το Γενικό Γραμματέα. Κύριε Τάραντ, σύντομα παρακαλώ. 15 δευτερόλεπτα λέει ο κύριος Τάραντ. Εγώ δέχομαι τις απόψεις του Γενικού Γραμματέα αν δεν γίνουν νέες ρυθμίσεις σε σχέση με το... Ε, με το ότι το μπαρ των βουλευτών θα γίνει μπαρ καπνιστών. Κοιτάξτε, για το θέμα α, ανάμεσα στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο ας κάνουμε όποιο είναι το αποτέλεσμα του σημερινού βραδινού αγώνα. Λοιπόν, να κερδίσει ο καλύτερος, λέει ο πρόεδρος, εγώ βλέπω ότι ο τελικός από ό,τι φαίνεται θα είναι εντελώς ευρωπαϊκός. Α, δυστυχώς έχουμε καθυστερήσει και ζητώ συγγνώμη από τους εκπρόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης που θα μας μιλήσουν για την α, κτηριακή τους πολιτική ο κύριος Μάρκ Σελινό από ε, το ΟΗΜΠΕ, ο κύριος Μπεκέ από το ΙΕΛ του Λουξεμβούργου και ο κύριος Ντουκέλ από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έχετε τρία λεπτά ο καθένας για μια σύντομη, μα πολύ σύντομη παρέμβαση. Ο κύριος Σέλινο. Όχι, ο κύριος Μπεκέ, αν επιτρέψετε, θα ξεκινήσει. Λοιπόν, ε, να σας ενημερώσω για δύο θέματα σχετικά με το Λουξεμβούργο. Το πρώτο αφορά το Ζωμονέ 2, που διαδέχεται το παλαιό κτίριο Ζωμονέ. Πρόκειται για ένα κτίριο 180.000 τετραγωνικών μέτρων, 3.700 άτομα χωρητικότητα με το σύνολο των υπηρεσιών της Επιτροπής στο Λουξεμβούργο. Θα μας δοθεί σε δύο στάδια το κτίριο, θα παραδοθεί σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο θα είναι για 2.700 υπαλλήλους από το Φεβρουάριο του 2023 ενώ η δεύτερη φάση από το Φεβρουάριο του 2024 θα φιλοξενήσει χίλιους επιπλέον συναδέλφους. Το κόστος είναι γνωστό από τότε που η αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή συμφώνησε το 2013. Δεν θα αναφερθώ ξανά στους αριθμούς. Να σημειώσω όμως ότι αποφασίσαμε να μην κτίσουμε επίσης και το κέντρο υπολογισμού γιατί εγκαταστάθηκαν εκτός κτιρίου σε άλλες κτιριακές υποδομές και ότι επίσης αντιμετωπίσαμε κάποιες απαιτήσει στον τομέα ασφάλειας πάρα πολύ σημαντικές που μας υποχρέωσαν να επανεξετάσουμε στοιχεία του κτιρίου στη σχεδίασή του και την οικοδόμησή του. Ξεκονομήσαμε κάποια χρήματα σε κάποιες πλευρές, είχαμε και επιπλέον χρήματα όμως ανάγκη, ε, συνολικά 17 εκατομμύρια επιπλέον. Δηλαδή ε, υπερβαίνουμε κατά 17 εκατομμύρια, 4% συνολικά την αύξηση και αύξηση της ε, χωρητικότητας του κτηρίου κατά 20%. Λοιπόν, αύξηση του προσωπικού, απλοποίηση της πρόσωψης, ε, κατάργηση μείον 6 και μείον 7 λόγω της αναθεώρησης της τοπικής νομοθεσίας σχετικά με τις θέσεις ε, στάθμευσης, μη κατασκευή ε, του κέντρου υπολογισμών και εφαρμογή νέων μέτρων ασφαλείας που μας υποχρεώνουν να καλύψουμε και το 35% των υπόγειων εγκαταστάσεων, κάτι το οποίο θα κοστίσει 21 εκατομμύρια. Υποβάλλουμε ένα σημείο μας στην αρχή επί του προϋπολογισμού, να μας επιτρέψει την αύξηση αυτή, εξηγώντας αναλυτικά όλες τις αλλαγές οι οποίες έχουν επισυμβεί. Ένα άλλο θέμα, για το οποίο θα είμαι πολύ σύντομος επίσης, πρόκειται για ένα κτίριο ε, για, για το κέντρο δημοσιεύσεων στο Λουξεμβούργο. Το κτίριο βρίσκεται στο τέλος της ζωής του, ο ιδιοκτήτης του θα το ε, καταστρέψει ουσιαστικά. Ε, και έχουμε μία προσφορά από την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου για να βρεθεί μία λύση η οποία θα μας επιτρέψει και να μείνουμε λίγα χρόνια επιπλέον στο κτίριο, αναβάλλοντας δηλαδή την αλλαγή και να νοικιάσουμε μετά ένα κτίριο το οποίο ε, είναι πολύ κοντά και το οποίο παρέχει λίγο μεγαλύτερη χωρητικότητα και με κόστος αρκετά ενδιαφέρον γιατί το κτίριο το οποίο νοικιάζουμε τώρα και λίγιο που να είναι το συμβόλαιο εδώ και 20 χρόνια τον νοικιάζουμε βέβαια και έχουμε υπογράψει το συμβόλαιο, το να νοικιάσουμε τις ίδιες επιφάνειες θα κοστίσει στην ίδια περιοχή 60% επιπλέον. Η ενδιάμεση λύση μέχρι τον Νοέμβριο του 2022 κοστίζει 35% επιπλέον και η τελική ε, κατάληξη της διαδικασίας αυτής μετά από τον Νοέμβριο το 2022 θα κοστίζει μόνο 20% επιπλέον και θα είναι πιο ευνοϊκή λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπεκέ. Ε, σημαίνει ότι μιλήσατε και για τον κύριο Σελινό. Ελπίζω όχι, λέει ο κύριος Μπέκε, Ο κύριος Σελινό λοιπόν να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ. Αν μου δώσει το τηλεχειριστήριο ο κύριος Μπέκε. Σύντομα λοιπόν οι τέσσερις βασικοί άξονες ε, με τους οποίους αναπτύσσει την κτηριακή της Στρατηγική Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναδιαπραγμάτευση για κάποιες συμβάσεις όταν η κατάσταση των κτηρίων το επιτρέπει και βρισκόμαστε στο προσδόκιμο ζωής. Αξιολόγηση της αξίας ε, της ε, περιουσίας που εμείς κατέχουμε με ανακαινήσεις και αναδιαρρυθμίσεις νέα κτίρια, αν τυχόν δεν μπορέσουμε να βρούμε λύσεις με τα δύο προηγούμενα και ε, εξορθολογισμός και ορθή χρήση του συνόλου των κτίριων. Τα βασικά κτίρια τα οποία έχουμε μπροστά μας είναι η εκμετάλλευση αν θέλετε του ε, L130 που θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε κατά 90.000 τετραγωνικά μέτρα την επιφάνεια σε δύο φάσεις, μία φάση που ξεκινάει από το 2015, 25 συγγνώμη, και μία δεύτερη από 25 μέχρι 30 που πρέπει να, για να πετύχει να αγοράσουμε και τα κτίρια Λουά 78 και Λουά 82. Ξέρετε ότι τελείγει και η σύμβαση για τον Μπορσέτ και υπάρχουν και αλλαγέ σε σχέση με τον Μπολιού και τα BU 29, 31 και 33 που είμαστε ιδιοκτήτες, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει οικονομικά. Το Μπρέντελ και Μπρέντελ 2 θα ανακαινιστούν. Οι ανάγκες μας σε επίπεδο επιφανειών χρήσιμων όπως δημοσιεύθηκαν την προηγούμενη άνοιξη είναι 80 με 150 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα για την περίοδο 2020-2024 για να αντακαταστήσουμε και τα κτίρια για τα οποία δεν θα μπορέσουμε να συνάψουμε ενδιαφέρουσες νέες συμβάσεις. Ε, δεν θα καθυστερήσω τώρα πάνω στο L130, έχει ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός βρισκόμαστε στα πλαίσια της πρώτης φάσης των εργασιών της Επιτροπής Επιλογής και τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 19. Αυτό ε, γίνεται ε, στα πλαίσια ενός διεθνούς φυσικά διαγωνισμού. Λοιπόν, σχεδόν 200.000 ε, τετραγωνικά μέτρα, αν συγκρίνουμε με τα 90 που έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα το κέντρο διασκέψεων θα αντικαταστήσει το Μπορσέτ και θα μας βοηθήσει στην αύξηση και επίσης ε, ε, εξελίσσεται η διαγωνιστική διαδικασία, δεν έχει ολοκληρωθεί και ένα τελευταίο σημείο θα δώσω το λόγο ε, στον υπεύθυνο θεμάτων ασφαλείας για την δημιουργία ενός κτηρίου υποδοχής στον Περλεμό. Ευχαριστώ. Το όνομα μου είναι Νικολάς Θα είμαι πολύ σύντομος για τα σχέδια για το κέντρο υποδοχής. Ο στόχος του κέντρου αυτό είναι να εξοικοποιήσει τους συνθήκες ασφάλειας για τους ε, επισκέπτες στον Περλεμόν ώστε να αποτρέψει τη χρήση όπλων. Έχουμε ανοιχτές μετάλλων αυτή τη στιγμή και ανοιχτές ε, συσκευές εντός του κτηρίου. Θα ήταν καλύτερα αν όλα αυτά λαμβάνουν χώρα εκτός του κτηρίου που θα είναι ε, προσαρτημένο στο κτίριο Μπερλαμό. Μερικά λόγια για τον Περλαμό. Το κέντρο υποδοχή θα είναι στην Εσπλανάντ, στην ε, Λεωφόρο Σαρλεμάνι. Άρα αυτοί που θα έρχονται από το μετρό θα παίρνουν ένα badge πρόσβαση στο κέντρο υποδοχή και μετά θα χρησιμοποιούν αυτό το μπάτζ για να μπουν στο κέντρο υποδοχή όπου θα αναλαμβάνει χώρα ο έλεγχο για να περάσουν συνέχεια ε, μέσα στο κτίριο η Εσπλανάδα ανάμεσα στο κέντρο θα είναι αποκλειστικά για οχήματα VIP και θα υπάρχει μια νέα είσοδος για τους VIP κατευθείαν από, την... από τον προάβλιο χώρο. Το χρονοδιάγραμμα το Ιούνιο του προηγούμενου ε, πήραμε άδεια σχεδιασμού. Υποβάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο ε, Γραφείο ε, Κοινοποίησεων το συμβόλαιο. Θα εκδοθεί στην επίσημη εφημερίδα στι επόμενε μέρε. Οι προσφορές θα ληφθούν στις αρχές του Νοεμβρίου, όπου θα γίνει και η επίσημη υποβολή στην αρχή προπολογισμού και αναμένουμε ότι θέλει δυνατόν να συνάψουμε σύμβαση ε, στα μέσα Φεβρουαρίου ανάλογα με την έγκριση. Μετά από μια προκατακτική μελέτη, οι εργασίες θα ξεκινήσουν τον Μάιο του, 2000, του 2019 και θα κρατήσουν 10 μήνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ε, διευκρινήσεις αυτές. Ε, Ζητώ συγγνώμη που σας πιέζω. Ο κύριος Ντουκέν από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την αντίστοιχη Υπηρεσία ε, Κτηρίων και ε, σας ευχαριστώ. Ο Γενικός Γραμματέας μας ενέκρινε σχέδιο δράσης για να βελτιώσουμε τα κτίρια μετά από τις συστάσεις ε, του ελεκτικού συνεδρίου. Για πρώτη φορά έχουμε προτεραιότητες σε σχέση με τη γεωγραφική υπηρεσία ε, για να αυξήσουμε τα κτίρια μας, ε, με τα κράτη-μέλη ε, να έχουμε συμμετοχή, να δούμε τι γίνεται με τα κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται και τις εγκαταστάσεις και να βελτιώσουμε την στέγαση. Εστιάζουμε στην υγεία και την ασφάλεια, στο περιβάλλον και την προβολή και την ε, δημοσιότητα. Δύο λόγια για τις βελτιώσεις και τον τρόπο που εργαζόμαστε. Για πρώτη φορά έχουμε διεύθυνση που συνεργάζεται με την ασφάλεια και τις υποδομές όπως σε διάφορα κράτη-μέλη. Έχουμε επιπλέον ανθρωπίνους πόρους από το 2018. Ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο για την υποστήριξη. Έχουμε εσωτερική λήψη αποφάσεων με διαφορετικό τρόπο ε, και ναι, βελτίωση στο λογισμικό μας. Ε, πώς επεκτείνεται το δίκτυο. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ε, ε ανοίγουμε στο Τουρκμενιστάν, Παναμά, Μογγολία, Κουβέιτ και υπάρχει το καθόδε ζήτημα της παρουσίας μας στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, όπου θα, ε, έχουμε παρουσία το 2019 στο Λονδίνο και κλείσαμε τα γραφεία μας στις νήσους Ολομόντα και ε, στην Τεχεράνη που μας φιλοξενούσαν οι Ολλανδοί. Είχαμε ένα γραφείο που χρησιμοποιούσαμε εκεί. Ε, μετακομίζουμε από τον Πελιάρ 100 και έχουμε και το project το τη Νέο ε, που έχετε δει στα πλαίσια της δημοσιονομικής διαδικασίας. Επίσης θέλουμε να αγοράσουμε στην Ουάσιγκτον γραφεία και σημαντικά ε, σχέδια έχουμε για το Κόσοβο, Νότια Αφρική, Ινδία, Ιράκ, Αφγανιστά, Κίνα και πολλά ακόμα κράτη. Ευχαριστώ. Ζητήσαμε από την κυρία Μόνικα Χολμάιερ να ε, μιλήσει. Θέλετε τώρα να μιλήσατε. Είναι ένα συμπίλημα ολόκληρο, οπότε ε, είναι συναρπαστικό τώρα να αντιδράσει κανείς ε, θερμό. Για το κτίριο Ζαμονέ, ναι. πώς έχει το κόστος. Είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο που είχαμε αποφασίσει στην αρχή. Και άρα και το νέο κόστος ε, είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει εμείς να αποφασίσουμε ως Επιτροπή Προϋπολογισμών. Γιατί σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό πραγματικά είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Έχω και άλλη ερώτηση για το κόστος εξοπλισμού του data center. 20 εκατομμύρια είχαμε μετά 21 εκατομμύρια και τώρα τίποτα μια παύλα. Τι είναι αυτή η παύλα και τι σημαίνει ακριβώς. Έχει καταργηθεί το κέντρο αυτό, data center, ε, ε, είναι πιο ακριβό, μετασκευάζεται, έχει εξαφανιστεί. Πού είναι το ποσό και τι έχει γίνει αυτό το κτίριο τελικώς. Και το, όπως και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλω να προειδοποιήσω για τις εξελίξεις ε, δεν ε, τις καταλαβαίνω πάρα πολύ ούτε εγώ που είμαι ε, η συγγήτρια ούτε η σκιώδης θα πρέπει για να μπορέσουμε να δουλέψουμε εγκαίρως να μας δίνετε στοιχεία και ποσά εγώ ως εισηγήτρια δεν μπορώ να διαμαρτυρηθώ ότι έχω την ενημέρωση πολύ νωρίς τελευταία στιγμή μου το χώνουν κάτω από τη μύτη μου και προσπαθώ να ενημερώσω τους χιώδης ηγητές για οτιδήποτε μαθαίνω και πραγματικά έχει αρχίσει και με εκνευρίζει σοβαρά αυτό, για να το πω έτσι, γιατί ε, είναι δύσκολο να ρωτήσεις, να διερευνήσεις κάποια στοιχεία και έχουμε την αίσθηση ότι είναι σκεμμένη αυτή η καθυστέρηση στην ενημέρωση για να μην χώνουν τη μύτη τους οι ε, καταλαβαίνω ότι γίνονται και κάποιες αλλαγές, αλλά στο κτίριο Ζάμονε το είπα και εγκαίρως ότι θα πρέπει νωρί να μας ενημερώνετε, εγκαίρως να συζητάτε μαζί μας και επίση εγκαίρως να μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Για το κτίριο ΛΟΑ 130 θέλω να πω ότι κομψά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να βάλει την έγκριση μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2019 ε, μας κοροϊδεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ποιος νομίζετε ότι θα συνεδριάζει Μάιο με Ιούλιο του 2019 εδώ σε αυτό το κτίριο. Τι θα έρθουμε νομίζετε για να αποφασίσουμε ειδικά για το νέο σας συνεδριακό κέντρο. Τι προγραμματισμός είναι αυτός. Έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά γίνονται από πρόθεση. Όλοι ξέρουν ότι του χρόνου έχουμε ευρωεκλογέ και Μάιο με Ιούλιο δεν συνεδριάζει ψυχή εδώ πέρα. Εντάξει, μπορεί για τον προπολογισμό να συνεδριάσουμε, αλλά ουσιαστικά αυτό είναι ανέκδοτο που λέτε. Ένα κύριο ε, που έχουμε εκατοντάδε εκατομμύρια να αποφασίσουμε, θα τα αποφασίσουμε, λέτε, από το Μάιο μέχρι τον Ιούλιο του 19. Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσω. Εγώ περιμένω το Μάρτιο να αποφασίσουμε και να το συζητήσουμε. Δεν γίνεται ε, να πέφτει πάνω στην αλλαγή της θητείας και πάνω σε ευρωεκλογές κάτι τέτοιο και το έχουμε ξανασυνδεί πολλές φορές και μετά χαλάμε τις καρδιές μας. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο 2019 είναι, για να το πω έτσι ε, κάπως εύσχημα, απολύτως no-go σε καμία περίπτωση και ελπίζω να έρθει νωρίς για να έχουμε τουλάχιστον την ευκαιρία τουλάχιστον να το σκεφτούμε για να μην πω για να το αποφασίσουμε και να μην ε, ε, ληφθούν ε, αποφάσεις ερήμην μας ή λόγω απουσίας μας αυτόματα να ελπίζουν κάποιοι ότι θα δοθεί έγκριση επειδή θα έρθουν τελευταία στιγμή. Κατά τα άλλα, χαίρομαι που έχουμε τώρα μια γενική εικόνα, μια επισκόπηση, ακόμα και είναι δύσκολη για τους συναδέλφους και τόσο μικρή, γιατί δεν γνωρίζουν όλοι το ιστορικό. Ήταν πολύ σύντομη παρουσίαση σήμερα. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, όλοι ο Πρόεδρος σκιώδη ηγητές, αναπληρωτές, η κυρία Γουαρδία Σάμπαλ δεν θέλει το λόγο. Εγώ, γιατί βλέπω ότι έχετε διάφορα έργα και, σχέδια και εξαγορά στην Ουάσιγκτον, στο Κόσοβο, Νότια Αφρική, Ιράκ, Αφγανιστάν, Κίνα, Ινδία κλπ. Δεν κατάλαβα πολύ καλά ποια είναι η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα πρέπει να ετοιμάσουμε πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που να αποδεικνύει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Λέτε στο έγγραφο ότι θα αγοράσετε κτίρια. Θα συνενώσετε τις πρεσβείες των διαφόρων κρατών μελών για να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες οικονομίες. Γιατί τελικά καταλήγουμε να έχουμε 29 πρεσβείες σε πολλές χώρες και αυτό είναι ε, έτσι κάπως γελίο και δεν ε, ενισχύει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολίτων. Θα σας ξαναδώσω το λόγο και στους τρεις. Μια σύντομη παρουσίαση σας παρακαλώ πολύ απάντηση. Και θα το εκτιμήσουμε αν είστε σύντομοι. Ευχαριστώ. Ένα σημείο μόνο για το data center, το κέντρο υπολογισμών. Τι είναι αυτό. Ε, εδώ μιλούμε για το συγκεκριμένο χώρο στον οποίο ε, είχαμε προβλέψει αυτές τις εγκαταστάσεις ε, των υπολογιστών. Αυτά από το 2015 είναι αλλού, από τότε που φύγαμε από το Ζάμονε. Και επειδή καταργήθηκε αυτό το εμβαδόν, υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στον ίδιο το σχεδιασμό. Έχουμε μια σειρά ε, εγκαταστάσεων ε, που δεν χρησιμοποιούνται, τις εγκαταστάσεις ψήξης ας πούμε εννοώ ε, για τους υπολογιστές που δεν υπάρχουν γιατί δεν υπάρχουν υπολογιστές πια εκεί, εξού και η Παύλα. Έχει καταργηθεί αυτό, έχει εκλείψει. Από την άλλη έρχεται να προσθεθεί κόστος και θυμίζω τα ποσά της παρουσίασης ότι είναι και με την αριθμική αναπροσαρμογή σε σχέση με τα όσα είχαν κατατεθεί το 2013. Είναι πιο σύγχρονα. Αυτή είναι μια σύντομη εξήγηση. Η πληρέστερη θα σας υποβληθεί ε, μετά το καλοκαίρι γραπτός. Η κυρία Χόλμα, σύντομα κάτι ξέχασε. Έχω μπερδευτεί γιατί υπάρχουν τα έξοδα για το data center Δεν υπάρχει το κόστος για τον εξοπλισμό του data center καθόλου. Οι υπολογιστές έχουν φύγει, άρα το έχετε καταργήσει εκεί πέρα. Ναι, διαβάστε παρακαλώ, ναι. Ε, έχουν φύγει σε άλλα μέρη στο Λουξεμβούργο, σε άλλες εγκαταστάσεις ε, που και φιλοξενούνται εκεί. Και η Γενική Διεύθυνση ε, Πληροφορικής ε, νοικιάζει κτίρια εκεί 20 εκατομμύρια δεν είναι οι υπολογιστές οι ίδιοι, είναι τα μηχανήματα για να ψύχουν τους υπολογιστές και άλλες υποδομές και δεν χρειάζονται γιατί έχουν φύγει οι υπολογιστές εξού και δεν αναφέρεται εδώ το κόστος. Κύριε Σελινό. Κύριε Πρόεδρε. Σημειώνουμε την περίοδο no-go που ανέφερε η συγγήτρια ε, απλώ ο διάλογος αυτός είναι δυναμικός, είναι ανταγωνιστικός και το χρονοδιάγραμμα εδώ είναι απλώ ε, ενδεικτικό. Να το διορθώσετε, λέει ο Πρόεδρος, και να ικανοποιήσετε έτσι την εισηγητρία μας. Ο κύριος Ντουκέν. Ναι. Ε, δύο λόγια μόνο. Όλα αυτά τα έργα που σας παρουσιάζουμε δεν είναι αγορές κτηρίων. Υπάρχουν και πολλές ενοικιάσεις. Για την εξωτερική πολιτική κάνουμε μεγάλες προσπάθειες να μοιραζόμαστε τα κτίρια. Βεβαίως ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ ε, να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και αυτό καμιά φορά περιπλέκει το timing και το χρονοδιάγραμμα ε, γιατί έχουμε προβλήματα σε σχέση με το μέγεθος των κτηρίων, αλλά το μέγεθος, μάλλον το παράδειγμα της Ουάσιγκτον είναι ενδεικτικό και χαρακτηριστικό. Θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερα κτίρια και να συμμετέχουν και άλλοι εταίροι εκεί. Και η Ευρώπη να μιλάει με μια φωνή και η Ευρώπη επίσης να είναι και στο ίδιο κτίριο ολόκληρη. Ε, τα κράτη-μέλη δεν έχουν πάντα αυτή την πρόθεση εκδηλώσει. Όχι, αλλά το Κοινοβούλιο, λέει ο Πρόεδρος, να παρακινήσει και να παροτρύνει τα κράτη-μέλη. Εμεί είμαστε Επιτροπή Προπολογισμών και θα πρέπει να αποδείξουμε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αν λοιπόν από διπλωματική σκοπιά ε, στις πρωτεύουσε έχουμε χώρους για την Ευρώπη, καλό είναι και οι διάφορες πρεσβείες να ε, συγκεντρώνονται εκεί. Η κυρία Χόλμαγερ, όταν θα ψηφίσουμε για αυτό το θέμα, παρακαλώ να μας εξηγήσετε ε, με ακρίβεια γιατί αυτό το κόστος του data center ήταν μέσα. Και τώρα θέλω να μάθω τι πληρώνουμε για νίκαια. Γιατί δεν διάβασα ποτέ έγγραφο ε, για χώρους που νοικιάζουμε και για το μίστομα. Δεν έχω καμία πληροφόρηση γι' αυτά, ούτε ότι προέκυψε αλλαγή στον προγραμματισμό και στο σχεδιασμό για το συγκεκριμένο data center. Καλό θα ήταν και οι Λουξεμβούργοι να μάθουν ότι μπορείς και να διαβάζεις πληροφορίες. Υπάρχει αυτό. και επιλέγω ότι δεν, ε, μάλλον ε, υποθέτω ότι δεν επιλέγουμε και τα ακριβότερα οικόπεδα για να χτίσουμε. Σας ευχαριστώ και τους τρεις, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και θα μας διαβιβάσετε και τα έγγραφα, όχι σε εμά κυρίως, στην κυρία Χόλμαγε. Και τώρα με αρκετή καθυστέρηση και σας ζητώ συγγνώμη, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσε οι συζητήσεις, ε, καλωσορίζω τους εκπροσώπους των αποκεντρωμένων οργανισμών ε, που εκπροσωπούνται από τον εκτελεστικό διευθυντή της Frontex φέτος. Ε, ο Frontex ε, είναι και στην επικαιρότητα ως οργανισμός και στην καρδιά των συνεδριάσεων συνόδων κορυφής. Είναι ακτοφυλακή και σύνοροφυλακή, επικεφαλής ο κύριος Φαμπρίς Λεζερή, τον οποίο και καλωσορίζω. Τρεις άλλες ενότητες οργανισμών των συνοδεύων ε, από τη δικαιοσύνη, εσωτερικά, κοινωνικά θέματα και από το συντονισμό των οργανισμών. Καλωσορίζω και τους άλλους εκπροσώπους εδώ παρόντες και με τη συμφωνία του εισηγητού κύριου Γκάιερ θα δώσω το λόγο στον κύριο Λιζερή για 10 λεπτά και λίγο λιγότερο αν έχει την καλοσύνη γιατί καθυστερήσαμε πολύ και σας ζητώ συγγνώμη. Κύριε Γενικέ Δευτέρα, έχετε το λόγο. Euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την πρόσκληση που απευθύνατε στο δίκτυο του συνόλου των εξωτερικών υπηρεσιών της Ένωσης. Η πρακτική την οποία ακολουθούμε εδώ και καιρό την εκτιμούμε δεόντως και θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί πράγματι πιστεύουμε ότι οι συναντήσεις αυτές είναι χρήσιμες για την σωστή κατανόηση της λειτουργίας μας. Όπως βλέπετε, το σύνολο του δικτύου των εξωτερικών υπηρεσιών ποικίλει. Ο Ευρωπαίος Νομοθέτης έχει αποφασίσει ότι διαφορετικές υπηρεσίες ανταποκρίνονται στην εφαρμογή ορισμένων εξωτερικού τύπου, εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν και σε σχέση με το δίκτυο θεωρούμε ότι η κατανομή των δημοσιονομικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να γίνεται επί τη βάση μιας μελέτης κατά περίπτωση των αποστολών των αρμοδιοτήτων και του ρόλου της κάθε υπηρεσίας των προτεραιοτήτων και των επιμέρους αναγκών. Θα ήθελα τώρα να υπογραμμίσω κάποια από τα επιτεύγματα του δικτύου αυτού. Καταρχάς, την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για τη μείωση 5% επιβεβαιώθηκε ότι όλες οι υπηρεσίες που λειτουργούν με κανονική ταχύτητα έχουν προχωρήσει σε 8,5% μείωσης, περισσότερο δηλαδή από όλα τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πρέπει να υπογραμμίσουμε την προσπάθεια αυτή να υπογραμμίσω εξ ονόματος του δικτύου ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά στην κατανομή των δραστηριοτήτων και έχουμε υπολογίσει ότι έτσι καταφέραμε να, να εξοικονομήσουμε 10 εκατομμύρια ευρώ σε τετραετή περίοδο μοιράζοντας το ανθρώπινο δυναμικό. Παράδειγμα, Δημιουργήσαμε ε, ένα, μια ομάδα για την προκήρυξη των θέσεων που είναι διαθέσιμη και ορατή σε όλους τους πολίτες. Περνάω τώρα στο θέμα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Υπάρχει ένα θέμα, το θέμα των νέων χρηματοδοτήσεων. Οι υπηρεσίες που μετέχουν στο δίκτυο πιστεύουν ότι εκεί όπου είναι εφικτό οι υπηρεσίες θα πρέπει να διευρύνουν τους ιδίους πόρους τους μέσω τελών και επιβαρύνσεων όπου κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Δεν είναι εφικτό φυσικά αυτό σε όλους τους τομείς, αλλά εκεί που είναι εφικτό το δίκτυο θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια. Μια μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συστήνει την αξιολόγηση νέων τέτοιων δυνατοτήτων. Απαιτείται επίσης περισσότερη ευελιξία. Ο κανονισμός και ο δημοσιονομικός κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπουν περισσότερες bespoke λύσεις, κατά περίπτωση δηλαδή. Σαν παράδειγμα, διαχείριση επί τη βάση των επιδόσεων, και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση μια σφαιρική, ενιαία, ομοιόμορφη αξιολόγηση των υπηρεσιών. Θέλουμε να υπάρξει κατά περίπτωση έλεγχος. Πάντα στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Παρασκευή μόλις, όπως είχε συμφωνηθεί, μας έστειλαν μία πρόταση για το ε, κανονισμό πλαίσιο. Όπως φαντάζεστε το έγγραφο αυτό είναι περίπλοκο και ταυτόχρονα είναι καθοριστικό. Καθοριστικό για την σωστή διαχείριση του προϋπολογισμού και τη λειτουργία μας. Απαιτείται δυστυχώς περισσότερος χρόνος, πρέπει να το εξετάσουμε προσεκτικά και να μπορέσουμε να εκφράσουμε εξ του δικτύου κάποιες θέσεις οι οποίες να είναι τεκμηριωμένες. Αλλά πάντως, βασική στόχη για μια ακόμη φορά είναι το νομικό πλαίσιο να καλύπτει επιμέρους τις πραγματικότητες της κάθε α, εξωτερικής υπηρεσίας. Ο γενικός κανονισμός αυτός θα πρέπει να επιτρέπει την κατάθεση προτάσεων του δικτύου οι οποίες δεν μέχρι τώρα στάθηκε δυνατό να γίνουν δεκτές και να συμπεριληφθούν στο πολιετές δημοσιονομικό. Παραδείγματα, ευελιξία, δυνατότητα ανταπόκρισης σε μη προβλεπόμενα συμβάντα, σαν παράδειγμα αύξηση υποχρεωτική των αναγκών σε ανθρώπινους πόρους, κάτι το οποίο συνέβη στην τελευταία περίοδο στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων. Ε, ευέλικτη κατανομή των πιστώσεων σε επίπεδο ε, δημοσιονομικό. Επίσης θα θέλαμε να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ε, και αποδοτική μέθοδος εργασίας μείωσης διοικητικού άρθρους, πλούστευση των χρηματοπιστωτικών, χρηματοοικονομικών κανόνων και επίσης τίθεται και το θέμα όπως είπα των νέων πόρων αυτό σημαίνει πιθανώς την αναθεώρηση του ε, ιδρυτικού κανονισμού έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την έβρεση νέων πόρων. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε τους νέους αυτούς πόρους, αλλά το μήνυμά μας είναι κάτι τέτοιο να είναι εφικτό ε, σε επίπεδο νομικού πλαισίου. Θα μου επιτρέψετε τώρα να υπογραμμίσω κάποιες από τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας, κάποιες από τις προκλήσεις που είναι γνωστές στο Κοινοβούλιο. Καταρχάς, ε, ε, ο συντελεστής χαμηλής διόρθωσης, χαμηλού επίπεδου διορθώσεων, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα ε, στην συνέχεια λειτουργίας των υπηρεσιών. Δεν θα αναφερθώ σε κάθε υπηρεσία, αλλά όταν βλέπουμε ότι πάνω από το 15% του προσωπικού ε, προέρχεται από τη χώρα που φιλοξενεί την υπηρεσία, εκεί τίθεται ένα θέμα δεοντολογικό. Για το Brexit υπάρχει θέμα απώλειας εμπειρογνωμοσύνης και αυτό θέτει σε κίνδυνο την επιχειρησιακή συνέχεια. Διάλογος επίσης με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Έχει μεγάλη σημασία αυτό Θέλουμε να έχουμε στενή συνεργασία ανάμεσα στο δίκτυο και τα ευρωπαϊκά όργανα και ε, θεωρούμε ότι η διαοργανική ομάδα εργασίας υπαρίθμου 2 είναι κομβικό μέσο για να το πετύχουμε. Και γι' αυτό θέλω σαν δίκτυο να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα υπόλοιπα όργανα. Δεν θα συνεχίσω. Ναι. Εκ νέου εκφράζω την ε, αξιολόγησή μας τη θετική για την προσπάθεια που κάνετε και ελπίζω να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Λετζέρη. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συνοπτικός. Φάρκας, υπεύθυνο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής για τις αρχές που ασχολούνται με θέματα εποπτείας. Τέσσερα λεπτά. Αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας από την δημιουργία του ΙΣΑ το 2011. Έχουμε συμβάλει σε ένα σταθερό σύστημα και στον υποπτικό τομέα η Ευρώπη για την ασφάλεια και την απασχόληση, η ΕΣΜΑ, για τη χρηματονομική αγορά, για την προστασία των επενδύσεων και EBA για τις τράπεζες και τους ε, οργανισμούς πληρωμών. Από τη δημιουργία έχουμε προχωρήσει την εστίασή μας, έχουμε μετατοπίσει την εστίασή μας στην αρχή θέλουμε να δημιουργήσουμε χώρο και να κάνουμε ενιαία βίβλο ε, κανόνων, αλλά τώρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες με έναν ε, συνεκτικό τρόπο και να πετύχουμε ε, μια επιπτική σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργότερα σήμερα θα ψηφίσετε σε αυτή την Επιτροπή για τη γνωμοδότηση ε, για τις τρεις επιπτικές αρχές και σε αυτή την πρόταση υπάρχουν ε, πολύ χρήσιμες προτάσεις από εμάς να προσπαθήσουμε να βρούμε συνέργειες ανάμεσα στις τρεις υπηρεσίε. Προσπαθούμε να πετύχουμε, ε, προσπαθήσουμε και στο παρελθόν και μας ενθάρρυνε η πρότασή σας να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες για περισσότερες ε, συνέργειες. Ωστόσο, στην τρέχουσα κατάσταση και στην ε, δημοσιονομική κατάσταση, οι τρεις υπηρεσίες αντιμετωπίζουν κάποιες προκλήσεις ιδιαίτερα που έχουν να κάνουν με τους περιορισμούς ε, που έχουμε από τη διάρθρωση της χρηματοδότησης. Να αναφέρω κάποιες από τις νέες ε, περιοχές τις οποίες ε, εστιάζουμε αυτές τις μέρες. Κατά πρώτον θα κάνω λόγο για κάποιες τομεακές και κάποιες κοινέ ε, που αφορούν και τις τρεις εποπτικές αρχές όσον αφορά τις τομεακές. Η ΕΠΑ αυξάνει τις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει καταστάσεις ε, διασυνοριακών υποθέσεων. Ε, επίσης, θα της αντεθεί εντολή ε, να ασχοληθεί με τις ασφαλιστικές εταιρείε στην Ευρώπη και αυξάνει τις προσπάθειές της για την Πανευρωπαϊκή Σύνταξη που είναι μια ε, πρωτοβουλία αυτές τις μέρες. Η ΕΣΜΑ από την άλλη πλευρά ασχολείται με τις κινητές αξίες και θα έχει μεγαλύτερες αρμοδιότητες στον τομέα της εποπτείας ε, του CCP και στον τομέα της εποπτείας μια ευρωπαϊκά CCP, τα οποία είναι συστημικά ε, σημαντικά στην Ευρώπη. Υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της κεφαλαϊκής, ε, στο πρόγραμμα για ε, δράση της κεφαλικής αγοράς. Προετοιμάζουμε τρεις συμφωνίες που θα είναι το τελευταίο πακέτο που θα ολοκληρώνει την νομική μεταρρύθμιση και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίση έχουμε ε, αυξημένες ε, περιπτώσεις ε, διαμεσολάβησης. Επιπλέον, δημιουργούμε έναν κόμβο δεδομένων για πληροφορίες στον τομέα του e-banking. Υπάρχουν κοινέ προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Θα αναφέρω δύο ε, anti-money laundering, EML για την καταπολέμηση ε, των, της παράνομης ε, κεφαλαίων. Στο πλαίσιο του Brexit και τις ευρωπαϊκές αρχές ε, ενδιαφέρονται για θέματα οικονομικής αστάθειας και αντιμετωπίζουν διαφορετικά σενάρια Επίσης, οι προσπάθειες σύγκλησης είναι πολύ σημαντικές στο πλαίσιο του Brexit. καθώ αναμένετε να αποχωρήσει το Μέλλον Βασιλείο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να σας απευθύνω το λόγο και να τονίζω τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο πλαίσιο του τρέχοντος προπολογισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για που μας διαφωτίσατε. Ο Χουάν Μενέντες Βάλντες από το Eurofound, Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία για τη Βελτίωση των Συνθήκων Ζωής και Εργασίας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε. Είναι τιμή μου σήμερα που βρίσκομαι εδώ εκ μέρους ε, των ε, υπηρεσιών ε, όπως είναι η Σεντεφόπ, το Training Foundation στο Τωρίνο, η την ασφάλεια και την υγεία στο Μπιλμπάο και Eurofound που εδρεύει στο Δουβλίνο. Θα ήθελα να ευχαριστώ την Επιτροπή που εστιάζει την συζήτηση σε συγκεκριμένε τομεί, πολιτική, σε συγκεκριμένα κλάστερς, γιατί είναι δύσκολο να δούμε, να εξετάσουμε τον περιπολισμό ενός οργανισμού χωρίς να δούμε τον τομέα τον οποίο αφορά και να το δούμε σαν ολότητα και να το δούμε σαν ολότητα χωρίς να, ε, να λάβουμε υπόψη μας, υπόψη μας οι οργανισμοί μας συμβάλλουν ε, ε, στην δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασία, καλύτερων θετικών εργασία και πολιτικέ που θέλουν να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτοί το τομεί ε, το γραμμών προπολογισμού που έχουν να κάνουν με το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση κτλ. του Κοινωνικών ε, Δικαιωμάτων και οι υπηρεσίες θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το όργανο για την ε, εφαρμογή. Ο προπολογισμό έχει παγώσει από το 2013 και θα πρέπει να ε, παρέχουμε αντιστάθμιση για τον, για τον πληθωρισμό Πρέπει να προβούμε σε κάποιες πληρωμές, να μειώσουμε κατά 10% και όχι 5% τον προπολογισμό μας. Και τα τέσσερις υπηρεσίε έχουμε κάτω από 100 εργαζόμενους, σε κάποιες περιπτώσεις 50 εργαζόμενους, άρα η μείωση δεν κοστίζει και δεν έχει αντίκτυπο. Ε, αν σκεφτούμε κάτι θα ήταν αφελές. Επιπλέον η μείωση ε, μας ενθαρρύνει να πετύχουμε καλύτερη αποδοτικότητα. Ένα παράδειγμα είναι... Ένα ρωτό παράδειγμα είναι οι συντεφόπιοι Eurofound μαζί κατάφεραν να εξοικονομήσουν ένα εκατομμύριο και έχουμε ένα μνημόνιο κατανόηση τέσσερι υπηρεσίε με ένα ε, αριθμό δραστηριοτήτων στον οποίο συμμετέχουμε από κοινού σε τήσια βάση. Η εξοικονόμηση δεν ήταν ε, αρκετή ε, ώστε να αποφύγουμε περικοπές που επηρέασαν δραστηριότητε, όπω είναι το θεματολόγιο, το greening, αλλά και βασικές δραστηριότητες των υπηρεσιών επλήγησαν. Γιατί θα πρέπει να επιμηκύνουμε τον κύκλο, τον χρόνο που θα τηρήσουμε, το χρονοδιάγραμμα που θα τηρήσουμε, παρά τα αιτήματα των ενδιαφέροντων μερών, όπως είναι το Κοινοβούλιο. Έχουμε μειώσει στην DEFOP τα updates ε, άλλη υπηρεσία έχει μειώσει τα risk assessments ή τις εκστρατείες. Το 2019 ίσως βελτιωθούν τα πράγματα γιατί η πρόταση έχει... Έχουμε μία αύξηση κατά 2% εκτός από τις δεφόπ θα έχουμε ένα νέο μέλος στο European Labour Authority που δεν θα υπερκαλύπτει τις δραστηριότητες των άλλων ε, υπηρεσιών. Μπορεί ενδιάμεσα όμως να μας ε, ζητηθεί να παρέχουμε κάποιο είδους αντιστάθμιση για τη δημιουργία της νέας υπηρεσίας και έτσι να έχουμε και άλλες περικοπές. Αυτό θα επηρεάσει δραστικά Τις βασικές λειτουργίες άλλων οργανισμών. Επίσης, ε, η συνέχεια των ε, ερευνών θα πρέπει να σταματήσουν οι αισθητικές ε, μελέτες Θα ήθελα να επιστρέψω την προσοχή σας σε κάποια θέματα που αφορούν τον προπολογισμό του 2019, η ΣΕΝΤΕΦΟ έχει περικοπές 350.000 παρόλο που έχει συμμορφωθεί με το, έχει συμμορφωθεί με το πλαίσιο. Ε, σε άλλη υπηρεσία υπάρχουν θέματα με την πρόσληψη υπαλλήλων. Τώρα όμως ε, ξοδεύουμε ε, ένα και περισσότερα ε, χρήματα για έρευνε τι οποίε είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε. Γιατί ε, αναμένεται ε, να αναλάβουμε δράση. Αυτό σας το, το, το, το τονίζω όσον αφορά την αξία του έργου μας εμπιστευόμαστε και ε, για την αξία του έργου. Βασιζόμαστε σε εσά να εξετάσετε την γνωμοδότηση την Επιτροπή σας και εσείς αποφασίσετε ποιε θα είναι οι προτεραιότητε που θα δοθούν στον κοινωνικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι ε, στο να σας ε, παραδώσουμε τα πιθανά αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριος Λεζιαρή που θα ξαναμιλήσει, αλλά τώρα υπό την ιδιότητα ε, του εκτελεστικού διευθυντή της Frontex για τις οργανισμούς που έχουν να κάνουν με την δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. δικαιοσύνη, εσωτερικές υποθέσεις, δηλαδή όλες οι υπηρεσίες τις οποίες βλέπετε μπροστά σας. Έχουμε επίσης και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Αγγελίας που θα ξεκινήσει. Να υπογραμμίσω εδώ κάποια από τα επιτεύγματα της ομάδας αυτής για τις εσωτερικές υποθέσεις και τη δικαιοσύνη. Έχουμε καταρχάς ξεχωριστά σημεία στις συνθήκες που ορίζουν τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ελευθεριών, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Όλες αυτές οι εξωτερικές υπηρεσίες είναι στην ουσία το λειτουργικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις πολιτικές αυτές. Στα hot spot που δημιουργήθηκαν σαν παράδειγμα στην Ιταλία, στην Ελλάδα το 2015, ασχοληθήκαμε με θέματα μετανάστευσης και θέματα ασφαλείας στα εξωτερικά σύνορα. Εκεί η ΆΖΟ, η Frontex, η Europol, η Eurojust συνεργάστηκαν τόπου με τις εθνικές αρχές. Είχαμε και την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που γνωμοδότησε στα θέματά της και μπορούμε να πούμε γενικότερα ότι συνεργαστήκαμε έτσι ώστε να αναπτύξουμε κάποιες διαδικασίες με στόχο την σωστή διαχείριση των ατάκτων μεταναστών, αυτών που ζητούν άσυλο και συλλογή δεδομένων έτσι ώστε να εμπλουτιστούν οι φάκελοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε ποινικέ και άλλες υποθέσεις. ιδιαίτερα στον τομέα της αστυνομίας και της δικαστικής συνεργασίας. Η Europol και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Ναρκωτικά και τις Ναρκωτικές Ουσίες συνεργάζονται και δίδουν στρατηγικές αναλύσεις για τις αγορές των ναρκωτικών ουσιών και το μέγεθος των απειλών. Και μια συλλογική τελικά προσπάθεια επίτευγμα είναι η ομάδα υψηλού επίπεδου για συστήματα πληροφορικής και διαλειτουργικότητα. Δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2016 και μπορεί να προσφέρει πολλά και σε επίπεδο ΕΑΖΟ, Ιουλίζα, Europol και η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για να προετοιμαθεί το νομοθετικό πακέτο σε σχέση με την διαλειτουργικότητα των υποθέσεων δικαιοσύνης και εσωτερικών δεδομένων και της τράπεζες δεδομένων που τις τεκμηριώνουν. Σχετικά με τον προϋπολογισμό τώρα, το 1 τέταρτο του προϋπολογισμού του τρίτου τμήματος αναφέρεται σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, 900 εκατομμύρια ευρώ. Παρά την αύξηση, οι υπηρεσίες αυτές ε, έχουν προχωρήσει στο 5% μείωση, έχουν ε, Τώρα όλες μαζί γύρω στους 2.000 υπαλλήλους. Δεν έχει υπάρξει μια ε, ισότιμη κατανομή των μειώσεων. Να πω ότι κάθε, περιουσία, κάθε εξωτερική υπηρεσία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ξεχωριστό τρόπο. Ε, όχι μόνο οι υπηρεσίες των οποίων διευρύνεται η εντολή, αλλά και οι υπηρεσίες οι οποίες διατάσσονται ουσιαστικά να αυξήσουν τις υπηρεσίες τους και ποσοτικά και ποιοτικά. Τώρα κάποιες προβλέψεις από το 19 και μετά. Η ομάδα των εξωτερικών υπηρεσιών στα θέματα αυτά θα προχωρήσει ακόμα την διαλειτουργικότητα των συστημάτων σαν παράδειγμα το αίτιας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα φέρει σε πολύ καλύτερη επαφή την EU-LISA, τη Frontex, τη Europol και τη Eurojust. Και θα χρειαστούμε επίσης και τη συμμετοχή της ΕΠΟΛ για να εκπαιδεύσει σωστά τους ε, υπεύθυνου ε, στα στελέχη που θα ασχοληθούν με την Τράπεζα Δεδομένων Αίτιας. Να πω ότι για το ΕΓΚΕ ε, το δίκτυο δηλαδή. Υπάρχουν πολλά που μένει να γίνουν στον τομέα της ψηφιοποίησης στους τομείς που καλύπτει το δίκτυο. Ε, σαν παράδειγμα, ανακατανομή των αριθμητικών στοιχείων έτσι ώστε να ελεγχθεί καλύτερα η επίπτωση της ε, κυβερνητικής, της, της, της βίας που ασκείται μέσω του διαδικτύου κτλ. Υπάρχει επίσης και το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου, σύστημα εξυγχρονιστικό για το Schengen και εδώ η Ιούλειζα και το Europol συνεργάζονται. Επίσης και το οργανωμένο έγκλημα και η υπηρεσία στη Europol ε, και η ένισα θα συνεργάζονται για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και τη βελτίωση των συνθήκων ασφαλείας και να υπογραμμίσω επίσης και τη δημιουργία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα σε συνεργασία με την Eurojust και την Europol που θα διευκολύνει την σωστή εφαρμογή των δραστηριοτήτων όλων των υπηρεσιών. Συνεργαζόμαστε επίσης και με γειτονικέ χώρες και εδώ θέλω να κλείσω και να σας ευχαριστήσω Πρόεδρε σας και τα μέλη σας για την προσοχή σας. Ελπίζω να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε στις απορίες σας. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά για την ενημέρωση αυτή. 20 λεπτά τώρα ερωτήσεις. Μπορεί η ψηφοφορία αντί για τις 11 και 4 να αρχίσει 11.30. Ο Hans Γκάιερ, ο μόνιμος ε, εισηγητής μας, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους Γενικούς Διευθυντές για τη σύντομη επισκόπηση των εργασιών των οργανισμών που ε, είμαι σε θέση να γνωρίζω είναι πολύ ευρύτερη λειτουργία από τη σύντομη παρουσίαση που έγινε. Χαίρομαι που ήρθατε σήμερα το πρωί στην Επιτροπή μας για να μας παρουσιάσετε ε, τα προβλήματα που έχετε, τις προκλήσεις ε, της αλλά και τις διοικητικές και τις οικονομικές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας και για μένα προσωπικά. Είμαι περήφανο που είμαι μόνιμο ηγητής για του εξωτερικού οργανισμού, αλλά στην Επιτροπή μα εδώ οι συνάδελφοι έχουν την τάση καμιά φορά, με εξαίρεση του σκιώδη που με ελέγχουν, οι περισσότεροι συνάδελφοι λένε ότι καλά έχουμε του ειδικού μα για του οργανισμού, α επιφορτιστούν εκείνοι να τα διεκπαιρώσουν και εμεί ασχολούμαστε με τα πολύ μεγάλα δημοσιονομικά ζητήματα. Και αυτό κατανοητό είναι. Αλλά είναι καλή ευκαιρία που έχουμε να τα ακούμε και να συζητούμε εδώ αυτά τα θέματα. Να δούμε ποιες αλληλεξαρτήσεις υπάρχουν ε, ανάμεσα στα πολιτικά ζητήματα που συζητούμε και την εκτέλεσή τους. Γιατί σημαίνει για σας. Ε, έχουμε καλή επαφή και ανταλλαγές ε, τακτά χρονικά διαστήματα. Έχω την ευκαιρία να επισκέπτομαι τους οργανισμούς αυτούς και με χαρά το κάνω. Ταξιδεύω ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιοδία και χαίρομαι να, που μπορώ να είμαι παρόν και όταν συνεδριάζει το δίκτυό σας για να διατηρούμε το διάλογο. Αυτό που με ενδιαφέρει σήμερα το πρωί κυρίως είναι τα εξής δύο να πω και να ε, <laughs> ζητήσω και την υποστήριξη της Επιτροπής μας. Στο προηγούμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, στο Μεσοπρόθεσμο, ορισμένα κράτη-μέλη τελικά κατάφεραν να συμφωνήσουν όταν προτάθηκε γενική περικοπή 5% του προσωπικού και των πόρων. Για να μπορέσουν διάφοροι ηγέτες να γυρίσουν στο σπίτι τους και να προβάλλουν ότι κόβουν το κεφάλι της λενέας γραφειοκρατικής ίδρας της Βρυξέλλες. Αν δούμε στην πράξη τι σημαίνει αυτό όμως και στις λεπτομέρειες, είναι δραματική η κατάσταση σε κάθε προπολογισμό του Κοινοβουλίου αγωνιζόμαστε και ακούω από τη γραμματεία του Συμβουλίου ότι δεν έχουν ομάδες μεταφραστών που να δουλεύουν παράλληλα δύο ομάδες και να μεταφράζουν ε, για να συνεδριάζουν οι ομάδες εργασίας του Συμβουλίου όπως θα επιδημούσα. Και έχει δραματική συνέπειες και στους δικούς σας οργανισμούς και είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Γιατί δεν έπρεπε κάθε οργανισμός μόνο να κόψει 5%. Όχι. Ταυτόχρονα ε, είχαμε και νέους οργανισμούς και νέα καθήκοντα και υπήρχε και μια ε, ομάδα μετατάξεων, αυτό το redeployment pool, ε, που πρέπει να στέλνουν εκεί προσωπικό, που δεν είναι 5% λοιπόν και ο κύριος Λεζερή μίλησε για το γεγονός ότι όλοι έχουν καλύψει το 5%, ορισμένοι οργανισμοί μέχρι και 9%. Και σε μικρούς οργανισμούς τέτοια περικοπή προσωπικού είναι οδυνηρή γιατί 5% του προσωπικού μπορεί να είναι λίγο σε κεφάλια, αλλά είναι πολύ σε πραγματογνωμοσύνη και σε καθήκοντα αποφασιστικά. Αυτό λοιπόν που έχω βάλει ως στόχο και στην ετήσια διαδικασία του προπολογισμού, αλλά και στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι αυτή η ανοησία που είναι συμβολική ε, πολιτική κίνηση και δεν ε, λύνει προβλήματα, να αποτρέπεται. Ένα άλλο που θέλω να αναφέρω σύντομα είναι η κατάσταση των εσόδων. Διαπληκτίζομαι πολλές φορές εδώ στην Επιτροπή για να βελτιωθεί αυτό. Δεξιά και αριστερά έχουμε ένα μπούσουλα για να συνεννοούμαστε. Ορισμένοι ανησυχούν μήπως κάποιος οργανισμός ε, που είναι υπερβολικά εξαρτημένος από τέλη που εισπράττει κινδυνεύει να μεροληπτεί. Δηλαδή μήπως πλησιάζει πάρα πολύ τους ενδιαφερόμενους από τους οποίους εισπράττει και πώς δεν μπορεί να διαφυλάξει την ανεξαρτησία της. Μια άλλη ομάδα βουλευτών έχει γενικά προβλήματα με τέλη και εισφορές και αύξηση και, γενικά επιβολή τέτοιων τελών και τα θεωρεί επικίνδυνα. Εμείς Προσπαθούμε να κινηθούμε ανάμεσα σε αυτές τις κόκκινες γραμμές το ΜΑ και το ΔΕ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και από οικονομίες. Και κοιτάξαμε και πού βρίσκονται τα όρια αυτών. Έγινε μια μελέτη ε, που ε, είχε πολλές συνεντεύξεις και με, με δικού σας Και απέδειξαν αυτές οι μελέτες ότι έχουμε εξαντλήσει τα όρια μας. 3-3% υπάρχει ως περιθώριο που δεν είναι και τεράστιο ποσοστό. Εγώ θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω και για την κατάσταση των εισόδων. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις και ευχαριστώ τους συναδέλφους που τις έκαναν. Δηλαδή, το ύψος των εσόδων δεν θα πρέπει να προσανατολίζεται στο διοικητικό κόστος διεκπαιρέωσης, δηλαδή να μην αφορούν τα τέλη την κάλυψη αποκλειστικά του διοικητικού κόστους, αλλά να δούμε και τι γίνεται με την είσοδο στην αγορά. Ε, όταν κάποιος παίρνει μια άδεια, ας πούμε, στην Αυστραλία. αυτό αυξάνει τα έσοδα του ενδιαφερόμενου που του δίνει στην άδεια, αλλά θα πρέπει αντίστοιχα να αυξάνει και το τέλος που καλείται να καταβάλει στον οργανισμό. Ξέρω όμως ότι διαμαρτύρονται κάποιε πολιτικές ομάδες εδώ. Θα ήθελα να το συζητήσουμε μαζί αυτό το θέμα με εσά. Πώς το βλέπετε, ποια είναι η δική σα εκτίμηση. Ε, είναι μια πρόταση της Deloitte αυτή. Καλά, το έργο δεν τελειώνει ποτέ, το δίκτυο διευρύνεται και οι προκλήσεις και τα καθήκοντα για τους οργανισμούς. Ακούστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ήδη από σήμερα, ακόμα και αν είναι στα σπάργανα αυτή η προσπάθεια και θα αρχίσει να λειτουργεί σε λίγα χρόνια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήδη από τώρα απομιζά χρήματα και προσωπικό από άλλους οργανισμούς για να στελεχωθεί και να βοηθηθεί να ορθοποδήσει. Και επειδή η ζωή είναι αυτή που είναι, όταν το πάπλωμα δεν φτάνει και το τραβάς μέχρι ε, το πρόσωπο, κρυώνουν τα πόδια και όταν το τραβάς πιο κάτω σε πονάει ο λαιμό σου. Δηλαδή τώρα παίρνουν λεφτά και χρήματα από τη Europol την ίδια για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Και στην προηγούμενη δημοσιονομική συζήτηση ε, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τους οργανισμούς που έχουν να κάνουν με ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας των κινδύνων κτλ. Και, και την Ευρωπόλ να την ενισχύσουμε. Οπότε δεν μπορούμε να το δεχτούμε ούτε στη δική μας επιτροπή να γίνονται τέτοιες κινήσεις. Να ενισχύονται οι οργανισμοί και διάφορες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τη δίωξη και την εσωτερική ασφάλεια. Αλλά αυτά δεν μπορούν να είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, παίρνει από τον ένα και τα δίνει στον άλλον αναγκαστικά, λες και είναι νόμος της φύσης. Θα πρέπει ε, ε, να πω ότι είμαι πολύ δυσαρεστημένος από αυτή την τακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω να μπορέσουμε να τη διορθώσουμε στην Επιτροπή μας. Το επόμενο που θα έρθει μπροστά μας είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Επασχόληση το European Labour Authority και θα πρέπει να έχουμε στεναρή στάση, να πούμε ότι μάλιστα θέλουμε τον οργανισμό αυτό να κάνει τη δουλειά του, να αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, αλλά γι' αυτό χρειάζεται το κατάλληλο προσωπικό και τους κατάλληλους ε, πόρους οικονομικούς. Και παρακαλώ μην τα πάρετε από κάπου αλλού τώρα, από κάποιον άλλο οργανισμό, που μπορεί αυτή τη στιγμή να μην είναι ε, ε, το φω τη δημοσιοτητα. αλλά και αυτοί κάνουν πολύτιμη δουλειά και του χρειάζονται αυτού και δεν θα πρέπει να περικόψουμε. Ο κύριος Μενέντες ε, Βάλντες τα είπε όλα αυτά πολύ ε, ευγενικά και εύσχημα ότι είναι αρνητική προτεραιότητα. Λοιπόν, θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα της επάρκειας των εσόδων να το δούμε ε, και στο διοργανικό διάλογο, αν χρειάζεται, για να παραμείνουν ομάδες εργασίας που αυτό τον καιρό δεν έχουν δουλειά. Και παρακαλώ τους οργανισμούς να μας στείλουν τις θέσεις τους ως προς την παρουσία τους. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να είναι παρόντες οι οργανισμοί καθ' όλη τη διάρκεια ε, μιας ομάδας εργασίας. Αλλά ε, τα δύο άλλα θεσμικά όργανα δεν θα το επέτρεπαν ποτέ κάτι τέτοιο για διάφορους λόγους δικούς τους. Οπότε η όλα ή τίποτα που είναι η σημερινή θέση των οργανισμών μου φαίνεται κάπως προβληματική θέση. Παρακαλώ να το ξανασκεφτείτε. Ε, εγώ θεωρώ ότι μπορώ να επιχειρηματολογήσω. Έχω αυτή την ε, εντύπωση ε, αλλά να είναι παρόντες εκπρόσωποι των οργανισμών στην αρχή της ενεδρίασης και να παρουσιάζουν τις θέσεις τους. Δεν θέλω να το απεμπολίσουμε. Θα δώσω το λόγο τώρα στους συναδέλφους. Ξέρω ότι θα είναι σύντομη. Ε, ο κύριος Όρμπριχτ. Μια παρατήρηση για τον Γιένς είναι πολύ σαφές ότι το έχει συνηθίσει αλλά και κάποιος από μας αποτελεί έκπληξη ότι η ερώτηση που θέτουν οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών είναι ευρωπαϊκή ή όχι. Μιλάνε για τους θεσμούς και για τις υπηρεσίες τους από όλους στην Ευρώπη από τους πολίτες. Η είναι, είναι ευρωπαϊκοί φορείς. Άρα δεν είναι αυτό το ερώτημα το είναι το πώς φερόμαστε στους φορείς αυτούς τους οργανισμούς. Είναι εργαλεία για τη δημιουργία πολιτικής, είναι αναξάρτητοι οργανισμοί. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για τη Frontex. Μιλάμε για τις νέες προτεραιότητες και για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Η προστασία των συνόρων προτεραιότητα το σύστημα ασύλου. Όταν ζητάμε λοιπόν τον προπολογισμό, θα πρέπει να έχουμε υπόψη. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες προς άλλες επιτροπές. Θα... Αν έχουμε διαφωνίες, ποιες θα είναι οι συνέπειες είναι οι πολιτικέ αυτέ έτοιμες, έχουν αποφασίσει ήδη τα μέλη για την προστασία των συνόρων. Ποια είναι η θέση της Frontex, ποιος είναι ο ρόλο τη Frontex γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην συγκεκριμένη ομάδα, έχουμε ξεκάθαρη πολιτική. άλλε υπηρεσίε, άλλοι οργανισμοί βρίσκονται σε αναμονή. Αυτά είναι βασικά. Πώ λοιπόν θα συζητήσουμε τον προπολογισμό αν δεν ξέρουμε ποιε είναι οι πολιτικέ. Και έχω υποψίσει ότι ακόμα και οι ίδιοι οι οργανισμοί δεν γνωρίζουν ποιε είναι οι πολιτικέ. Άρα, πώ μπορούμε να στήσουμε τον προπολογισμό όταν δεν είμαστε σαφεί. Γιατί θυμάμαι. Θυμάμαι ένα κείμενο που αφορούσε 100.000 άτομα. 50.000 πόσους θα χρησιμοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Θα πρέπει να είμαστε πιο σαφείς. Αν θέλουμε να συζητήσουμε λοιπόν για τον προπολογισμό, θα πρέπει να έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη κατάσταση ω προ την πολιτική που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Και τα δύο και οι οργανισμοί. Άρα δεν έχει να κάνει με τη Frontex. Θα πρέπει να ε, είμαστε σαφείς ως προς ε, θα πρέπει να υπάρχει μια ενότητα, να μην κάνουμε διαχωρισμό ανάμεσα στις ε, αποκεντρωμένες υπηρεσίε και στα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των υπηρεσιών για τις παρουσιάσεις τους και θα επικεντρωθώ στις ε, εποπτικές αρχές. Πολύ σημαντικός ο ρόλος τους, ώστε να ε, υπάρχει ορθή ρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών. Όσον αφορά την οικονομική σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι προϋπόθεση για την ε, οικονομική ολοκλήρωση και την γυρότητα ε, της αγοράς. Υπάρχουν δυστυχώς τρεις υπηρεσίες εντός της ομάδας, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και η ΕΣΜΑ. Θα ήθελα να, ρωτήσω κάποια, να θέσω κάποια ερωτήματα. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα είναι να υποστηρίξουν τους ε, εθνικούς επόπτες ώστε να έχουν υψηλής ποιότητας εποπτεία. Ποια είναι η αποδοτικότητα σε περίπτωση παραβιάσεων. Σε πολλές περιπτώσεις τα συνταξιδετικά ε, ταμεία ε, έχουν θέματα με τους κινδύνους που υπάρχουν σε σχέση με την σταθερότητα την οικονομική του συνταξιδετικού τομέα κατά πόσο ακολουθείτε τις ε, εξελίξεις, ε, τις τεχνολογικές για να μειώσετε ε, το ρίσκο στις χρηματοδοτικές αγορές, ποια είναι η θετικότητα του τραπεζικού συστήματος. Και τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορείτε να μας πληροφορήσετε περισσότερο για την υποστήριξη που παρέχεται στις εθνικές αρχές εποπτείας στη διαδικασία του stress testing των τραπεζών. Ευχαριστώ κύριε Χολμάια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να υποστηρίξω στεναρά τον κύριο Γκάιερ. σε ό,τι αφορά ε, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη, τους οργανισμούς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλλον όχι, θα αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένα στατικό τρόπο. Ε, αν δεν υπάρχουν νέα καθήκοντα και νέες υποχρεώσεις, τις ε, αγνοεί. Ε, και όταν τις αποφασίζει, εντάξει, και το Συμβούλιο Επίσης δεν έχει σωστή στάση. Η παράτυπη μετανάστευση δεν είναι κάτι που έχουμε ορίσει εμείς ως καθήκον νέων, ούτε η τρομοκρατία και η ασφάλεια. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, οπότε δεν χρειάζεται στατική αντιμετώπιση, αλλά δυναμική αντιμετώπιση. Δεν είναι ε, κάτι που έχει να κάνει ε, με τις επιθυμίες μας για το πώς φανταζόμαστε τον κόσμο. Οι ανάγκες προκύπτουν ε, από τις δυναμικές εξελίξεις. Τώρα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν μέχρι το 2020 να έχουν 10.000 ε, ε, υπαλλήλου στείλει στη Frontex. Πολύ φιλόδοξο αυτό και πολύ σπορτίφ για να δούμε αν θα το πετύχουν. Αυτές οι δυναμικές λοιπόν αποφάσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων δεν ακολουθούνται ε, από την εξίσου δυναμική αντιμετώπιση της Κομισιόν, αλλά τη στατική αντιμετώπιση της Κομισιόν που τους δίνει ένα εκατομμύριο. Και στο παρελθόν χρειαζόταν αύξηση επικοδότηση. Τα ίδια ισχύουν και για Eurojust, Europol και για να είμαι και για την EU Liza. Αλλά το βρίσκω εξίσου θλιβερό αυτό που κάνει το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο συζητάει και για ψήφισμα και για ό,τι άλλο θέλετε, αλλά το Συμβούλιο κατά αρχήν αρνείται τη συζήτηση γιατί δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Θα πρέπει να κοιτάξουμε όμως ποιες είναι οι ανάγκες, ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τι απαιτούμε από τους οργανισμούς. Και όχι ποιες είναι οι επιθυμίες και οι προθέσεις του καθενός για τον προϋπολογισμό. Καλό είναι να είμαστε φιδωλοί στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και τακτοποιημένοι, αλλά να μην αντιμετωπίζουμε με τέτοιο παράλογο τρόπο, για να το πω έτσι, τις υπηρεσίες αυτές και τους οργανισμούς. Ευχαριστώ, κύριε Στουπχέ. Σύντομα, κύριε Πρόεδρε, διότι συμφωνώ τόσο με τα όσα είπαν οι προλαλήσαντες. Κύριε Λιτζερή, έχω μια παρατήρηση. Σας εκτιμώ πάρα πολύ και σας σέβομαι, αλλά μας έχετε στείλει ένα έγγραφο για τους οργανισμούς δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων και εδώ υπάρχει μια φρασούλα που λέει και δίνει την εντύπωση ότι λυπάται γι' αυτό ότι η αύξηση των πόρων δεν εφαρμόστηκε με τρόπο ανάλογο ε, μεταξύ των διαφόρων οργανισμών. Και εκπλήσουμε λίγο έτσι αντικειμενικά. Ε, λες και ήσασταν εσείς συνδικαλιστής του οργανισμού ή των οργανισμών και καλείστε να ε, υπερασπιστείτε τα συμφέροντα όλων των οργανισμών. Ο δικός μας στόχος ποιο είναι. Οι οργανισμοί αυτοί να παίρνουν ε, τα μέτρα και τις δυνατότητες που ανταποκρίνονται στις πρωτοβουλίε και τις προτεραιότητε πολιτικής που εμεί του αναθέτουμε και στα θέματα των εσωτερικών και της δικαιοσύνης, τα είπε η Μόνικα Χολμάγερ. Αν θέλει η Frontex να έχει 10.000 επιπλέον σύνοριοφύλακες να προσλάβει, ε, η υπηρεσία της Λισαβόνας που παρατηρηθεί την τοξικομανία και, τα ναρκωτικά δεν χρειάζεται αντίστοιχη αύξηση και ανάλογη. Ε, για το λόγο αυτό, συμφωνώ με τους συναδέλφου, θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνουμε υπόψη κάθε φορά τι επιχειρησιακές προτεραιότητες και αντίστοιχα να δίνουμε τα απαραίτητα μέσα. Το Συμβούλιο αποφασίζει και η Επιτροπή εκτελεί. Στο Γιουλάιζα τώρα έχουμε εγκρίνει μια σειρά νέων νομικών βάσεων για τις τράπεζες δεδομένων. Εσείς τα ξέρετε αυτά καλύτερα. Ε, Eurodac, Etias και τα διάφορα άλλα. Ε, αυτό είναι μεγάλη δουλειά για τον εξυγχρονισμό της πληροφορικής. Άρα είναι φυσιολογικό να δοθούν εκεί περισσότερα μέσα και κονδύλια. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν ε, ήδη αποφασιστεί. Έχουμε τη νομική βάση. Θα ήθελα να συμφωνήσουμε γι' αυτό, σας παρακαλώ. Καλή ήσυχη μεταχείριση μεταξύ των οργανισμών, αλλά δεν έχει νόημα. Κατανοώ τη δυσκολία του ρόλου σας, γιατί μιλήσατε και ε, εξ ονόματος οργανισμών σε κάποιο συγκεκριμένο κλάδο, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω για την πλήρη ισότητα εδώ. Ε, δεν έχει δει κανένα άλλο το λόγο. Θα ήθελα να απευθυνθώ εγώ στον κύριο Μενέντες Βαλντές, γιατί η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης είναι κάτι το οποίο θα κυριαρχήσει στο μέλλον. Από την έννοια αυτή θα ήθελα λίγο να μας διαφωτίσετε ρώτησε και ο Γιάννης Γκάιερ, τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Αρχή Απασχόλησης, Labor Authority. Πρόσφατα είδαμε τη συζήτηση για το καθεστώς των οδηγών φορτηγών και είδαμε πόσο δύσκολο είναι να συγκλίνουμε στην Ευρώπη. Για την ανεργία, νομίζω, ο ε, ε, οργανισμός ΣΕΝΤΕΦΟΠ, τον οποίο εκπροσωπείται, ασχολείται με αυτό το θέμα και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πιο σαφείς προτάσεις και πιο δεσμευτικές ε, για τις μεταρρυθμίσεις που προτείνονται για την καταπολέμηση της ανεργίας ιδιαίτερα των νέων. Θα ήθελα να εκφράσω μια ευχή να είμαστε πιο εχμηροί και πιο ε, στεναρεί στις προτάσεις μας ε, για νέα προγράμματα, ας πούμε, επαγγελματικής κατάρτισης των νέων, τώρα που σχεδιάζουμε και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ορισμένες μελέτες χρειάζεται να είναι πιο εχμηρές για να ε, στραφούμε στο μέλλον. Θα σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις πάρα πολύ σύντομα, μοιραία και με την αντίστοιχη απογοήτευση. Άρα θα το ξαναπούμε. Πρώτος, για να απαντήσει ο κύριος Φάρκας. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Έχω, έχω τέσσερα ερωτήματα. Θα τα απαντήσω ανάποδα. Το πρώτο, τελευταίο μάλλον, ήταν ε, ότι υπάρχει EBA στις ε, εθνικές αρχές ως προς το trust testing. Η EBA κάνει ένα ευρωπαϊκό stress test ε, κάθε τρία χρόνια, μεθοδολογία αυτού του stress test και όλη η άσκηση είναι εκτή σε όλες τις αρχές. Υπάρχει δημόσια διαβούλευση και οποιαδήποτε αρχή που θέλει να κάνει stress test πέρα από το δείγμα το οποίο προτείνει η EBA που είναι 50 τράπεζε σε όλη την Ευρώπη. Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για την εφαρμογή της μεθοδολογίας για άλλε τράπεζες. Οι εθνικέ αρχές επιλέγουν ε, να εφαρμόσουν τα ίδια στάνταρ. Επιπλέον έχουμε ένα σετ ε, οδηγιών, διευθυντήριων γραμμών και ενθαρρύνουμε τις αρχές να τις εφαρμόσουν αυτές τις ε, κατευθυντήριες γραμμές όταν αποφασίζουν να διεξάγουν δικό τους stress τεστ. Η τρίτη ερώτηση έχει να κάνει με την τεχνολογία και οι τρεις αρχές είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με ένα σχέδιο δράσης στη FinTech με δύο στόχους. Ο ένας είναι να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν στι νέε τεχνολογικέ εξελίξει στον ε, χρηματοοικονομικό τομέα και θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ε, οικονομική ολοκλήρωση και να δημιουργήσουν μια ενιαία αγορά σε διάφορου τομεί, όπω είναι οι πληρωμέ και άλλε υπηρεσίε. Άρα κοιτάμε τι ευκαιρίε και πώ μπορούν ε, οι ρυθμιστικέ αρχέ και οι εποπτικέ αρχέ να ενθαρρύνουν τη χρήση αυτών των ευκαιριών. Από την άλλη πλευρά μελετάμε του κινδύνου που προκύπτουν από την καινοτομία στην τεχνολογία όπως είναι το κυβέρνο, κυβέρνο επιθέσεις. Ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ πλοκό θέμα γιατί δεν ε, συμπεριλαμβάνει μόνο τις οπτικές αρχές αλλά και άλλες υπηρεσίες με άλλες αρμοδιότητες. Το δεύτερο ερώτημα που με ρωτήσατε έχει να κάνει με τα συντεξιτικά συστήματα για τις επενδυτικές πολιτικές. Η ΕΟΠΑ δεν ε, εποπτεύει μονομένα συντεξιτικά συστήματα ταμεία, αλλά τις αρχές που είναι υπεύθυνε για την εποπτεία και χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για να διασφαλίσουν ε, ότι οι εποπτικές αρχές εφαρμόζουν ε, ε, τους κανόνες που αφορούν τα συνταξιδικά ταμεία όσον αφορά το χρηματιστήριο αξιών αυτό που είναι σημαντικό είναι να ε, συγκρατείτε εντό του πλαισίου επενδύσεων ώστε να μην ε, τεθείτε σε κίνδυνο οι συντάξει. Η πρώτη ερώτηση, τι υποστήριξη παρέχουν ε, οι υποπτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Αρχές στις εθνικές αρχές. Έχουμε ήπια εργαλεία όπως είναι καθητήριες γραμμές, έχουμε ε, αξιολογήσεις, ε, peer reviews, έχουμε μελέτες, αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων των αρχών, αλλά σε ένα πιο ε, αυστηρό πλαίσιο υπάρχει και διαμεσολάβηση σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Με την εφαρμογή αυτών των εργαλείων προσπαθούμε να υπάρχει συμμόρφωση και συνέπεια. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τομέων. Όπως γνωρίζουμε υπάρχει μια νέα οπτική αρχή στον τραπεζικό τομέα, ενώ στους άλλους τομείς. Ε, η ΕΣΜΑ έχει κάποιες οπτικές αρμοδιότητες. Ευχαριστώ. Merci. La parole est maintenant à monsieur. Ο κύριος Χουάν Μενέντες. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. για τις σχέσεις ανάμεσα στα θεσμικά όργανα και τις εξωτερικές υπηρεσίες. Εμείς δεν είμαστε ευρωπαϊκά όργανα όπως τα υπόλοιπα, αλλά απαιτείται να υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση στις γραμμές τις οποίες ακολουθούμε και είναι σαφές ότι θα πρέπει κάθε τομεακή κοινοβουλευτική επιτροπή ε, να ε, έρχεται σε επαφή απευθείας με τις εξωτερικές υπηρεσίες και έτσι θα έχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες το ταχύτερο δυνατόν. Τώρα βέβαια οι κοινοβουλευτικές επιτροπές θα πρέπει να καθορίσουν το επίπεδο προτεραιοτήτων να προβλέψουν επίσης ε, τους τρόπους με τους οποίους θα προωθήσουν τις πολιτικές τους που έχουν σαν στόχο την αύξηση του κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στις χώρες και με τις γειτονικές χώρες. Ο κύριος Ντεπρέ είπε ότι αν κάποιος αυξήσει την προτεραιότητα στα εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να μειώσει το επίπεδο αν θέλετε προσοχή στα εσωτερικά. Δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν σημαίνει ότι αν υπάρξει αύξηση του βαθμού προτεραιότητα σε ένα συγκεκριμένο κλάδο θα υπάρξει αντίστοιχα μείωση σε κάποιον άλλο. Ίσως εδώ να μην έχω καταλάβει κάτι σωστά τότε στην ερώτησή σας. Για το θέμα της κινητικότητας, η αρμόδια αρχή για θέματα εργασίας αναφέρθηκε σε αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε για δίκαιη κινητικότητα στην Ευρώπη, να δούμε ποια είναι η θετική και η αρνητική πλευρά. Λειτουργούμε συμπληρωματικά. Ασχολούμεθα με θέματα ανεργίας, με θέματα ανεργίας νέων, με θέματα βοήθειας στον τομέα της ανάπτυξης των ικανοτήτων και της κατάρτισης Νομίζω ότι στηρίζουμε έτσι, ε, μπορούμε να συνδράμουμε γενικότερα τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, ο κύριος Λετζερή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το αν η υπηρεσία γνωρίζει το ποια είναι η εντολή. Φυσικά ναι, έχουμε ένα ιδρυτικό κανονισμό, κάθε υπηρεσία εξωτερική έχει ένα ιδρυτικό κανονισμό Εμεί εδώ ασχολούμεθα, όπως είπα, με θέματα, με θέματα εσωτερικών υποθέσεων και θέματα δικαιοσύνης, ελευθεριών και αν μου ρωτήσετε να σας πω ποιος είναι ο ρόλος του Frontex είναι προφανώς να ενισχύσει τα εξωτερικά σύνορα για να διασφαλιστεί έτσι η εύρυθμη λειτουργία της κινητικότητας στο εσωτερικό της Ένωσης, στα εσωτερικά σύνορα. Θα συμφωνήσω επίσης λέγοντας ε, ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει μια στατική αντιμετώπιση ε, των δημοσιονομικών πόρων των υπηρεσιών. Σε ορισμένους τομείς βλέπουμε ότι σύμφωνα και με την εντολή την οποία έχουμε θα πρέπει να προετοιμαστούμε να προετοιμάσουμε δράσεις για να αποφύγουμε κάποιες κρίσεις. Αλλά αν συμβούν κάποιες κρίσεις τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της θα πρέπει να μπορέσει να αντιδράσει και οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι αρκετά ευελικτές έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν και να ενισχυθούν αν αυτό απαιτείται και να αναδιπλωθούν εκεί όπου χρειάζεται για να αντιμετωπίσουν τις κατεπίγουσες καταστάσεις. Σχετικά τώρα με το ότι η κατανομή των πόρων δεν έχει κατανεμηθεί δίκαια. Δεν έχει γίνει δίκαια. Τι εννοούμε με αυτό. Εννοούμε ότι υπάρχουν ε, αλληλοεξαρτήσεις ανάμεσα στις υπηρεσίες. Και από ό,τι φαίνεται ότι μέσω της ενίσχυσης ορισμένων υπηρεσιών όπως η Frontex, όπως η Europol, έμεσα αυτό δημιουργεί νέες αρμοδιότητες και νέα βάρη και για τις άλλες εξωτερικές υπηρεσίες. Όταν σαν παράδειγμα αρχίσαμε με μαζικό τρόπο να στέλνουμε στην Ιταλία και στην Ελλάδα συνοριοφύλακες, υπήρξε ανάγκη να συμμετέχουν και οι υπόλοιπες εξωτερικές υπηρεσίες έτσι ώστε να είναι οι ομόλογοι μας παρόντων, παρόντες για να ασχοληθούν με θέματα ετούντων ασύλου ή ε, με θέματα ποινικών διαδικασιών. Κύριε Πρόεδρε, έχω την αίσθηση ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις, αν ε, συμφωνείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος και τους τρεις, γιατί ήσασταν σαφείς και ε, συνοπτικοί όπως έπρεπε ο μόνιμος εισηγητής μας δεν θέλει να πάρει το λόγο για να κλείσει τη συζήτηση. Θα έχετε τη δυνατότητα να συναντηθείτε εκ νέου, έχετε δύσκολη αποστολή. Δεν είναι καθόλου εύκολο να ασχολείται κανείς με θέματα τα οποία εν πολύ είναι αντιφατικά. Απαιτείται να είναι κανείς ευέλικτος, απαιτείται να είναι ελαστικός και ε, θα έχετε όλοι μας τη στήριξη όταν προετοιμάσουμε το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας και ζητώ συγγνώμη για την πίεση χρόνου την οποία σας επιβάλαμε. Σας ευχαριστώ. Καλή επιστροφή στις υπηρεσίες σας. Θα συνεχίσουμε τώρα με τις ψηφοφορίες. Θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες με σημαντική καθυστέρηση και γι' αυτό ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους δεν ήμασταν αρκετά αποτελεσματικοί, αλλά έγιναν πολύ πλούσιες συζητήσεις σήμερα το πρωί και θα ήταν λάθος ίσως να μην αφήσουμε τους ομιλητές να εκφραστούν γιατί πράγματι μας διαφώτισαν επαρκώς. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, βάλτε σας παρακαλώ τις κάρτες σας στα μηχανήματα για την ηλεκτρονική ψηφοφορία για να κάνουμε μια δοκιμαστική. Αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Όχι. Δύο δεν ψηφίσατε. Πέρασε. Ωραία. 14 υπέρ, τρία κατά. Ό,τι και αν ψηφίζα. Λοιπόν, ψηφίζουμε την έκθεση του κύριου Γκάιερ. Κανονισμό για την τροποποίηση κανονισμών που θεσπίζουν ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και κανονισμό σχετικά με τι χρηματοοικονομικέ αγορέ. Η τροπολογία υπαριθμών 37 ψήφι υπέρ. Υπέρ. Αν είστε υπέρ, να σηκώσετε το χέρι σας παρακαλώ. Εγκρίνεται. Η ε, τροπολογία υπαριθμών 1 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμό 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμών 10 ψήφι Αμπλοκ, μήπως μπορούμε να τις ψηφίσουμε φωνές από κάτω. Α, que vous êtes euh, Συμφωνείτε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Αν δεν διαφωνεί κανείς. Ωραία. Κύριε Γκάιε, συμφωνείτε. από ποια τροπολογία μέχρι ποια τώρα όμως. Όλες, όλες. Όλες. Alors je les Κατά αποχές εγκρίνεται το σύνολο των τροπολογιών. Ε, τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε ονομαστικά. Αρχίζει τώρα. Θα ψηφίσατε όλοι. Ένας δεν ψηφίσε. Ακόμα. Α, τώρα εντάξει. Πέρασε. Εγκρίνεται. 21 ψήφοι υπέρ και 2 κατά. Τώρα, ο λόγος στο γενικό μας ηγητή, τον κύριο Μορεσάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα συνάδελφοι. Θα ψηφίσουμε δύο μεταφορές, αιτήσεις μεταφοράς, απόφαση 17 και 18. 31 ε, εκατομμύρια φορούν ε, από τη γραμμή MFE που δεν χρειάζεται ε, στην CFSP και DCI, στην ΚΕΠΑ δηλαδή. Γιατί εκτός από το MFA e με τη Γεωργία δεν υπάρχει πίστοση για τέτοια χώρα. Τα 20 εκατομμύρια για την ΕΠΑ προτείνω ως εξής. 6 εκατομμύρια να καλύψουν το κόστο ε, τη αποστολή εμφυλευτική στο Ιράκ. Έχω κάνει αντίστοιχε ερωτήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ποιο λόγο το χρειάζεται αυτό. Και η απάντηση είναι, λέει, διότι έχουν τους εξή δύο λόγους. Τα 14 ε, εκατομμύρια που είχαν ήταν για την περίοδο Οκτώβριο του 17 με Οκτώβριο του 18, άρα για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο χρειάζονται λεφτά και επίσης υπάρχει κάποιο επιπλέον κόστος ασφαλείας. για την αποστολή μας εκεί. Ε, άρα εκεί πηγαίνουν αυτά τα 6 εκατομμύρια. Το επόμενο είναι 5 εκατομμύρια ε, για μια νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιεμένη. Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να υποστηριχθεί ο μηχανισμός ε, του ΟΙΕ στο Τζιπουτί για να ε, περνούν προς την Ιεμένη απρόσκοπτα τα εμπορεύματα και αυτό είναι εντάξει καταρχήν, αλλά έχω μια μικρή τεχνική ερώτηση διευκρινιστική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί εγώ έχω κάνει γραπτέ ερωτήσει και στην απάντησή σα μου λέτε ότι 4,44 εκατομμύρια χρειάζεστε και τα υπόλοιπα 0,56 γιατί το έχετε στρογγυλέψει στα 5 εκατομμύρια. Εγώ ε, συνιστώ να υπερψηφιστεί αυτή η μεταφορά και τα υπόλοιπα 9 εκατομμύρια αφορούν τη μη διάδοση των πυρηνικών και τον αφοπλισμό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το λαθρεμπόριο όπλων ε, στην Αμερική και στις αραβικές χώρες. Αυτά είναι τα 20 εκατομμύρια. Είναι η πρώτη απόφαση ε, το 17 το 2018 να το ψηφίσουμε, αλλά γιατί ζητάτε 5 εκατομμύρια και όχι 4,44. Η δεύτερη της μεταφοράς 18 προτείνεται να μεταφερθούν 11,5 ε, εκατομμύρια από τη μακροοικονομική βοήθεια στο DCI για το Σαχέλ και το καταπίστευμα για την ασφάλεια και τα λοιπά, ε, για την καταπολέμηση της παράτυπης ε, μετανάστευσης και την αντιμετώπιση των εκτοπισμένων στην Αφρική. Και αυτό προτείνω να υπερψηφιστεί. Ωραία, να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί προτείνει 5 εκατομμύρια για την Ιεμένη. Ποιο θα απαντήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατά τα πρώτα, ευχαριστήσω τον κύριο Μουρισάν για την υποστήριξή του και για τι δύο προτάσει. Για να είμαι σύντομο όσον αφορά το ερώτημα του, πράγματι, από την στιγμή που υποβάλαμε την πρόταση για τη μεταφορά σε αυτήν την επιτροπή, υπήρξε μια επαναξιολόγηση των αναγκών ε, της αποστολής στην Ιεμένη και υπήρξε μια εξήμψη προς τα κάτω στα 4,44 ε, εκατομμύρια από 5 εκατομμύρια. Ωστόσο θα ζητήσω από την Επιτροπή αν είναι πρόθυμη να εγκρίνει την ε, μεταφορά όπως είναι. Προβλέπετε ότι ως το τέλος Ιουνίου για τον προπολογισμό ε, θα έχουμε κάποιες ε, ελλείψεις. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα στενά τους επόμενους μήνες και νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο όπως είναι αποστολές ε, στην στις Φιλιππίνες και στην, στην Κεντρική Δημοκρατία. Άρα έχουμε ένα πλεόνασμα 0,5 εκατομμυρίων που δεν θα χρειαστούν ε, στην ΙΕΜΕΝ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, σε αυτές τις νέες πρωτοβουλίες. Και ε, υπόσχομαι να κρατάω ενήμερο τον εισηγητή ως προς το τι θα γίνει με αυτά τα 0,5 εκατομμύρια. Ευχαριστώ πολύ. Για την ΕΠΑ, προσοχή, γιατί πέρσι πήραμε ε, αρκετά κονδύλια ε, τα αφαιρέσαμε και μετά από λίγους μήνες χρειάστηκε να την ξαναπροσθέσουμε. Η κυρία ε, Γκρέσλε, έχω μια ερώτηση για την αίτηση μεταφοράς 18 και ερωτώ πόσα χρήματα καθυστερούν τα κράτη-μέλη για το καταπιστευματικό ταμείο για την Αφρική. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γκρέσλα για την ερώτηση αυτή. Είναι γεγονός ότι οι ε, πληρωμές και το χρονοδιάγραμμα συμφωνήθηκε με τα κράτη-μέλη για να καταβάλουν ε, τις συνεισφορές τους στο καταπίστευμα για την Αφρική και μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν καθόλου καθυστερήσεις ως προς την καταβολή αυτών των ε, οφείλων. Και επίσης θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή 14% ε, των συνολικών ε, πληρωμών στο καταπίστευμα συνολικά ε, προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον όχι, διορθώνει ο μιλητής από άλλους δωρητές. Ε, πάντως τα κράτη-μέλη δεν έχουν καθυστερήσει αυτή τη στιγμή τις πληρωμές τους. Η κυρία Γκρέσλε. Κοιτάξτε, διάβασμα ξέρω, ανάγνωση δόξα το Θεώ καλά. Αυτές οι απαντήσεις που μας στείλατε είναι πάρα πολύ προβληματικές και ε, σάτυρα ουσιαστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να πληρώσουν. Το Συμβούλιο έρχεται να επικυρώσει αυτή την απέτηση και απευθύνεται στα κράτη-μέλη. Λοιπόν, ερωτώ. Πόσα χρήματα καθυστερούν τα κράτη-μέλη στο Trust Fund. Αυτό που μας διαβάσατε το διάβασα και εγώ. Και υπάρχει καθυστέρηση και αν δεν το γνωρίζετε ζητώ να αναβληθεί αυτή η μεταφορά γιατί δεν θα πρέπει εμείς να κάνουμε εδώ διάφορα πράγματα που δεν πατάνε στα πόδια τους. Αυτά τα κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε σωστές δουλειές και να ασκούμε και πίεση. Αυτά και ευχαριστώ. Ναι, αλλά αυτό το θέμα του καταπιστεύματος έτσι κι αλλιώ είναι λίγα τα λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βάζουμε πέντε δεκάρε και τα κράτη-μέλη βάζουν τα υπόλοιπα. Και υπάρχει μια κάποια αδράνεια στο σύστημα που φοβάμαι ότι κινδυνεύει να αναπτυχθεί. Λοιπόν, σύντομα, τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν υποχρεώσεις, αλλά από το Ταμείο δεν περνάνε. Ζητώ συγγνώμη, δεν είμαι βέβαιος αν κατάλαβα καλά. Πώς λέμε στην απάντησή μας ότι καθυστερούν τα κράτη-μέλη, τις πληρωμές τους. Αν θέλετε να συνενθώ διμερώς με την κυρία Γκρέσλε για να καταλάβω τι εννοεί. Μα όχι, μας ενδιαφέρει όλους αυτό το θέμα, δεν είναι της κυρίας Γκρέσλε. Ποιες είναι οι καθυστερήσεις των κρατών μελών ε, για να κάνουν τις πληρωμές τους ε, στο καταπιστευματικό ταμείο. Λοιπόν, Ας ε, το αφήσουμε εδώ. Αν θεωρεί ο Γενικός Συγητής ότι έχει ενημερωθεί επαρκώς, να ψηφίσουμε. Ο κύριος Μούρεσαν. Ναι, Πρόεδρε, αλλά αυτό που ρώτησε η Ίγκε Γκρέσλα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να μας απαντήσει αυτή τη στιγμή, εμεί δεν είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε με τη σειρά μας και δεν μπορούμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία, διότι ε, θα θεωρείται ε, ότι ψηφίστηκε αυτόματα. Εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ ή κατά αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να δώσει την πληροφόρηση που χρειάζονται οι συνάδελφοι. Θα πρέπει να καταψηφιστεί η αίτηση μεταφοράς και να την υποβάλει και πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θεωρείτε ότι μπορούμε να την υπερψηφίσουμε αργότερα κατά τη διάρκεια του έτους. Αργότερα πότε δηλαδή, το Σεπτέμβριο, κύριε Ρέλ. Um, thank you, Chair. I, I Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν μπορώ παρά να επαναλάβω ε, τα όσα γνωρίζω. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, δεν έχουν καθυστερήσει τα κράτη-μέλη να καταβάλουν τις πληρωμές τους. Από πού μάθατε εσείς ότι καθυστερούν τα κράτη-μέλη. Εγώ προσ... θα προσπαθήσω να το τσεκάρω και να επανέλθω αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχουν καθυστερήσεις ε, καταβολής πληρωμών από πλευράς κρατών μελών. Κυρία Κρέσλε. Εσείς που ξέρετε τις πληροφορίες, είναι σαφής. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν μιλάω τα καλύτερα αγγλικά, αλλά σας διαβάσω τι απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα αγγλικά. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά το 2017 ε, οι συνεισφορές των κρατών μελών και ανέρχονται στο 14%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν επιπλέον ε, επανειλημμένα. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του στις 28 Ιουνίου επανέλαβε αυτή την έκκληση. Τώρα τι μου λέτε ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει 82% και τα κράτη-μέλη μόνο 14%. Τι μου λέτε δηλαδή ότι 86% το πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη μόλις το 14%. Ε, παρακαλώ να μου απαντήσετε. Ζητώ συγγνώμη που δεν κατάλαβα την ερώτηση από την αρχή. Ε, στην παρούσα φάση πώς έχει η κατάσταση. Το 14% του συνόλου των πόρων των καταπατησματικών ταμείων προέρχονται από άλλες πηγές ε, πλην του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, EDF. Ε, έχουν συμφωνηθεί ε, χρονοδιαγράμματα για το 14% με τα κράτη-μέλη και γι' αυτό το 14% δεν υπάρχουν καθόλου καθυστερήσεις. Τα κράτη-μέλη σέβονται απολύτως τις υποχρεώσεις τους και τις δεσμεύσεις τους. Τούτων όλων λεχθέντων, επανειλημμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ότι έχουμε έλλειμμα χρηματοδότησης για το καταπιστευματικό ταμείο της Αφρικής και για τη Βόρεια Αφρική και για την υποσαχάρια Αφρική. Αυτό το θέμα συζητήθηκε και στο Συμβούλιο επί Μακρόν, όταν συζητούσαν τη δεύτερη δόση για τους πρόσφυγες και την καταβολή στην Τουρκία και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε συνέχεια και συμφώνησε για να κλείσει αυτό το έλλειμμα χρηματοδότησης για την υποσαχάρη Αφρική θα δοθούν επιπλέον 500 εκατομμύρια από τα κράτη-μέλη. Αυτά ακόμα δεν έχουν δοθεί. Είναι νέα δέσμευση που έχουν αλάβει τα κράτη-μέλη και δεν έχουν ανταποκριθεί αν υπάρχει καθυστέρηση εντό εισαγωγικών, αυτή έχει να κάνει με τη νέα ανάληψη υποχρεώσεων από τα κράτη-μέλη να ε, συνεισφέρουν επιπλέον 500 εκατομμύρια. Ζητώ συγγνώμη για τη σύγχυση, ελπίζω τώρα να έγινε σαφέ. Ζητώ συγγνώμη που ξαναπαίρνω το λόγο. Δεν καταλαβαίνω την ενημέρωση. Τι γράφεται εδώ πέρα. 602 εκατομμύρια έχουν συμφωνηθεί και 27 εκατομμύρια έχουν καταβληθεί. Και αυτά τα 27, πού θα τα θα ξύνουμε πάτους συρταριών από στον προϋπολογισμό. Αν δεν γνωρίζετε, να το δούμε το μεσημέρι. Αλλά με βάση αυτά που μας λέτε, εγώ δεν είμαι σε θέση να αποφασίσω. Έχω την αίσθηση ότι κάτι τρέχει που στρέφεται κατά του συμφέροντο και του κόσμου επιτόπου. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτή την τακτική. Κατ' εξαίρεση. Να ψηφίσουμε την υπόθεση αυτή το απόγευμα, γιατί συνεδριάζουμε το απόγευμα έτσι ώστε να έχουμε όλα τα διαθέσιμα. Συνεπώς λοιπόν βάζουμε στην άκρη το 17 θα πρέπει να αποφασίσουμε για το 18 τότε. Όχι, λάθος, λάθος λέει ο πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε το 17. Ηλεκτρονική κλίση. Ψηφίζεται. Ψηφίσατε όλοι. Δύο ψήφοι ακόμα. Πέρα της ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 2 κατά. Και το 18 θα ψηφιστεί ξεχωριστά το απόγευμα. Τι ώρα? Στο τέλος της συνεδρίασης για να έχουμε χρόνο τότε. Ανάμεσα στις 5 και τις 5.30. 5.30 λοιπόν. Εντάξει. Θα ακούσουμε τον κύριο Ashworth τώρα για τις υπόλοιπες μεταφορές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο μεταφορές, δύο αιτήσει μεταφορών και οι δύο προερχόμενες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 111 εκατομμύρια για την πρώιμη παιδική ηλικία. θα υπάρξει εξοικονόμηση χρημάτων και από τα θέματα αμοιβών, μιας και δεν έχει ακόμα διοριστεί ένας επιπλέον δικαστής. Ζητήθηκαν επίσης 185.000 για επιπλέον έκτακτο προσωπικό για τη δημοσίευση ε, νέων ε, νομικών αποφάσεων, δικαστικών αποφάσεων Μόνο σε συνοπτικό τρόπο βέβαια γίνεται αυτό και αυτό θα πρέπει λοιπόν να χρηματοδοτηθεί και από εξοικονόμηση της καθυστέρησης ε, έναρξης διαγωνιστικών διαδικασιών. Δεν υπάρχουν προβλήματα λοιπόν με τις μεταφορές αυτές, μπορούμε να τις εγκρίνουμε. Εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα για τις δύο αυτές μεταφορές και δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, γίνονται δεκτές. Ε, καλώς. Τώρα, κτηριακή πολιτική, Χολμαϊερ. Ευχαριστώ. Αρχικά, όσον αφορά το κτίριο της ΕΑΤ στο Παρίσι, βρίσκεται σε ένα κτίριο στο Λονδίνο προς το παρόν και εξαιτία ε, μιας γρήγορης αποφασής μεταφερθεί στο Παρίσι Πρέπει να βρούμε ένα κατάλληλο κτίριο. Θα παρακαλέσω την Επιτροπή να μας δώσει πληροφορίες σχετικά με... Δεν χρειάζεται να γίνει αυτό τώρα σε αυτή τη συνεδρίαση, αλλά το Σεπτέμβριο παρακαλώ. Τι γίνεται με τη μετακόμιση. Γιατί το κτίριο της ε, ΣΕΠΑ είναι νοικιασμένο μέχρι το 2020. Με την ΕΜΑ επίσης έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε μία ρήτρα ε, μετακόμιση το 2020. Θα πρέπει να πληρώσουμε πρόστιμο βέβαια. Θα πρέπει να έχουμε πιο σαφείς πληροφορίες. Το κτίριο τώρα έχει μια συνολική επιφάνεια 4.150. Το καινούργιο είναι πάνω 5.000. Άρα τα, τα έξοδα είναι πιο ε, χαμηλά στο Παρίσι από ό,τι στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο συνολικά είχαμε 3,7 εκατομμύρια το έτος στο καινούριο κτίριο 3 εκατομμύρια. Έχουμε περισσότερο χώρο, περισσότερη χώρο για τις συνεδριάσεις και χαμηλότερο ενίκιο. Μας βοήθησε και ε, η γαλλική κυβέρνηση με μια χρηματοδότηση 7 εκατομμυρίων και με αυτή τη χρηματοδότηση μειώνονται μειώνεται το ενίκιο. Επιπλέον 1,4 εκατομμύρια θα μας παρέχει η γαλλική κυβέρνηση. Θα ήθελα ε, να συγχαρώ ότι σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μπορούμε να βρούμε ένα, μια καλύτερη ευκαιρία ένα καλύτερο κτίριο από στο Λονδίνο. Έγινε πολύ καλή δουλειά και μας υποστηρίξει και η γαλλική κυβέρνηση. Δεν έχουμε λόγο να παραπονιόμαστε επομένω. Σας ευχαριστώ για την πλήρη απάντησή σας και γνωμοδότησή σας, κυρία Χόλμαγερ. Συνεπώς ψηφίζουμε ηλεκτρονική κλίση, παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. 18 υπέρ, μία κατά. Washington. Θα είμαι σύντομη και σε αυτό. Είμαστε σε ένα 11 όρφο κτίριο γραφείο. Θέλουμε να αγοράσουμε το κτίριο. Θα πρέπει να γίνει η αγορά αυτό το έτος των συνολικών εμβαδών είναι 12.887 τετραγωνικά μέτρα. Η ΑΕΔ έχει πάνω από 6.000 τετραγωνικά μέτρα. Τα υπόλοιπα ε, τα καταλαμβάνουν άλλοι οργανισμοί. και ε, πλέον τα τρονικά μέτρα παραχωρούνται σε πρεσβείες. 31 συνεργάτες συνολικά συστεγάζονται, ε, υπάρχουν 131. Ε, Υπάρχει χώρος στάθμευσης Υπάρχουν πλέον έξοδα στην αγορά, 2,2 εκατομμύρια. Είναι τα έξοδα για τους μεσίτες, τους δικηγόρους κτλ. Επιπλέον έξοδα για την ασφάλεια, 2 εκατομμύρια για την επίπλωση 1,4 εκατομμύρια, ανακαίνιση στα επόμενα 20 χρόνια 12,5 εκατομμύρια και για την διοίκηση έσοδα 17 ε, ε, εκατομμύρια από την επινοικίαση, 55 εκατομμύρια έσοδα Είναι θετική γενικά η εξέλιξη, θα υπάρξει συγχρηματοδότηση και θα ήθελα να έχουμε την έγκρισή σας γιατί είναι πολύ ε, λογική και πολύ συμφέρουσα η προσφορά. Σας ευχαριστώ για τη σύσταση αυτή, κύριος Δεπχέ. Ζητώ συγγνώμη, μια ερώτηση έχω γιατί δεν σας παρακολουθούν διερμηνείς με την ταχύτητα που διαβάζετε τα ποσά. Το συνολικό ποσό της εξαγοράς πόσο ήταν. Ποιο είναι το συνολικό ποσό ε, για την αγορά του κτίριου. Κύριε Χολμάγερ. Λοιπόν, συνολικό ε, κόστος όπως σας είπα και το τσέκαρα 102, μια στιγμή να το βρω. 9,65 και 13 εκατομμύρια ε, τόκοι ε, προστίθενται. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν 180 και κάτι ψηλά εκατομμύρια.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 98,4 ε, συν 13,575. 112 αντί για 102. Ήταν τυπογραφικό το λάθος αυτό. Τι είναι αυτό, ευρώ ή δολάρια. Ευρώ, ευρώ. Ευρώ. Όχι δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, Ζητώ συγγνώμη, εγώ θυμάμαι ε, ότι για μια εικοσαετία είναι πιο ακριβό. Είμαστε γύρω στα 180 εκατομμύρια, λέει ο κύριος Δεπρέ. Εγώ έχω 98 εκατομμύρια και 13 εκατομμύρια 575, τάδε τάδε φόρους. Ε, τόκους, συγγνώμη. 1,84% ε, είναι το επιτόκιο. Εντάξει, για 112 γράψαμε 102 κατά λάθο. Συγγνώμη. Κύριε Ντουκέν, μια που είστε ακόμα παρόν, πώς θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να διευκρινίσουμε κάτι. Σε δολάρια είναι η τιμή για την αγορά του, κυρίου, είναι, ε, του κτηρίου 104 εκατομμύρια δολάρια. 104 εκατομμύρια δολάρια. Βεβαίως σε ό,τι ε, αφορά το δικό μας προϋπολογισμό για να είναι ξεκάθαρα έχουμε μετατρέψει με την πιο πρόσφατη ισοτιμία τα δολάρια σε ευρώ. Βεβαίω, σε περίπτωση που δανειστούμε το σύνολο θα είναι πιο ψηλό το κόστος των τόκων. Αν ε, δανειστούμε λίγο λιγότερα από 104 εκατομμύρια μπορεί να είναι πιο χαμηλό το επιτόκιο. Η κατάσταση λοιπόν που σας ε, περιγράφει ε, δείχνει μία προσωμείωση που έχουμε κάνει με ε, τα σημερινά επιτόκια και τη σημερινή ισοτιμία. Και ποια είναι η διαφορά της τιμής αγοράς, της τιμής του σχεδίου με τις, τους τόκους και τη σημερινή ενοικίαση. Εγώ αυτό που σας διάβασα, λέει η κυρία Χόλμαγερ, αφορά το ευρώ και ισοτιμία 0,8597. Τα είπα σε ευρώ και δεν έχω τα στοιχεία ε, σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Συμπέρασμα λέει ο Πρόεδρος. Ε, δεν χρειάζεται να, ε, να θεωρήσουμε αυτή την ε, συναλλαγή. Τρέχει. Εσείς κυρία Χολμάγερ είστε θετική. Ωραία. Ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται 17 υπέρ 2 κατά. Κυρία Χολμάγερ, έχετε ακόμα το λόγο για την κτηριακή μας πολιτική. Υπάρχει ένα αίτημα από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για ένα κτίριο για το κτίριο Μπελιάρα 100 η υπηρεσία εξωτερική δράση θέλει να ε, παρατείνει ε, το διάστημα μίσθωση από μια τριετία σε μια εξαετία. Αυτά τα πήραμε την περασμένη Πέμπτη το βράδυ μετά το Στρασβούργο. Δεν τα έχουμε μελετήσει ούτε εγώ ούτε οι σκιώδει εισηγητέ. Εμεί δεν έχουμε πρόβλημα ούτε καμία αντίρρηση, αλλά θα προτείναμε να το θεωρήσουμε ενημέρωση τώρα και να αποφασίσουμε οριστικά το Σεπτέμβριο. Και να ρωτήσω κάτι γιατί δεν νοικιάσανε το κτίριο για έξι χρόνια από την αρχή, αλλά πρώτα για τρία συν τρία. Έτσι από περιέργεια ρωτώ, γιατί το βάλατε τρίτη, για να μην μπαίναμε τώρα σε αυτή την άσκηση. Ε, σύντομα, σύντομα, γιατί έχουμε μεγάλο θέμα που ακολουθεί. Θέλω να πω ότι ε, όταν υποβλήθηκε η πρόταση ε, πρόκειτο για μια αετή μίσθωση ε, και υπάρχει ελάχιστη περίοδος ασφαλείας που είναι τριετία και έγινε εξαετία. Αλλά η συνολική μίσθωση αφορά εννέα Αυτό είναι ένα θέμα εσωτερικής, κάτι μετασκευών που γίνονται εκεί που μας βγήκαν πιο ακριβές. Ωραία, να το κρίνουμε το Σεπτέμβριο, λέει ε, η κυρία Χολμάγερ, αλλά θεωρεί η υπηρεσία εξωτερική δράση ότι θα το εγκρίνουμε. Και το ίδιο για την αντιπροσωπεία στο Παρίσι. Το Παρίσι δεν χρειάζεται τώρα να το συζητήσουμε με την ησυχία μα το Σεπτέμβριο. Προτείνω να αναβληθεί το Παρίσι. Καλώς θα περάσουμε τώρα στη μελέτη που ζητήθηκε από την ε, ειδική υπηρεσία του Κοινοβουλίου για τις ε, επιδόσεις των διαφθρωτικών ταμείων υπό τη διεύθυνση του κυρίου Μπάκλα, του καθηγητή Μπάκλα του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης. Καλωσορίζω τους εμπειρογνώμονες λοιπόν του European Policy Research Center του, της Γλασκόβης και δίνω το λόγο στον, στους κυρίους Φάρι και Γκάλλα. Φάρη έχει το λόγο. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Να ζητήσω συγγνώμη γιατί ο κύριος Μπάτλερ δεν μπόρεσε να έρθει. Είμαι όμως με τον συναδελφό μου τον Φάιμπε Ιαγκάου. Η παρουσίαση μας βασίζεται από μία έρευνα από το EPRC την πολιτική ε, συνοχή ως προς την ε, χρηματοοικονομική της ε, απόδοση. Όσον αφορά τους στόχους, η έρευνά μας ήθελε να παρέχει μια γενική εικόνα για την κατάσταση, για την δημοσιονομική εκτέλεση του 2014 έως 2020 και να αναλύσει τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την εκτέλεση και να εξάγει κάποια συμπεράσματα για την πολιτική συνοχή στο πλαίσιο του πολιτικού δημοσιονομικού ε, πλαισίου για το 2020. Θα μοιραστούμε την παρουσίαση με τον Φάμπια. Θα δείξω το συνολικό pattern της πολιτικής συνοχής σε επίπεδο ε, κρατών μελών και προγράμματος. Μετά θα δω κάποια θέματα για να εστιάσω σε εξωτερικούς παράγοντες, κοινωνικό-οικονομικό Κόντεξ και μετά θα αναλάβει ο Φάμπια για να επεξηγήσει κάποιες στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπιστούν τα θέματα της εκτέλεσης και θα συνεχίσει με συμπέρασματα και συστάσεις. Η ανάλυση είναι πολύ επικίνδυνη για δύο λόγους, για πρακτικούς λόγους, γιατί μόλις περάσαμε το δεύτερο, περάσαμε στο δεύτερο μισό του προγράμματος για να δούμε πώς ε, προχωράει. Από το 7 στο 13 υπήρχαν θέματα απορρόφησης και γι' αυτό τώρα πλέον έχουν, υπάρχουν πιέσεις για ε, τις ε, αρχές προς την εκτέλεση. Η ανάλυση της χρηματοοικονομικής εκτέλεσης των πολιτικών συνοχής. Δόθηκε προσοχή σε ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκό επίπεδο, το ρυθμό α, των πληρωμών και επίσης είναι σαφές πόσο σημαντικό είναι τα θέματα που αφορούν την χρηματοοικονομική εκτέλεση από συγκεκριμένα κράτη-μέλη για να προετοιμάσουν ε, τις ε, ε, προτάσεις τους για μετά το 2020 έγινε ανάλυση δεδομένων, αλλά χρησιμοποιούμε και ε, ε, πληροφορίες από EPRC και το IQ Network από 15 κράτη-μέλη. Δημοσιονομική εκτέλεση. Έχουμε μια γενική εικόνα εδώ των πληρωμών και των υποχρεώσεων. Στον πρώτο πίνακα βλέπουμε τις ε, πληρωμές, την μπλε γραμμή. Δείχνει την απόδοση το 2007-2013 και η κόκκινη γραμμή την απόδοση ως, ε, που έχουμε μέχρι τώρα από το 2014 στο 2020. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ρυθμός πληρωμών είναι χαμηλότερο σε σχέση με το 2013. Το ποσοστό βλέπουμε των πιστώσεων είναι χαμηλότερες, ε, χαμηλότερος αριθμός των πληρωμών στα πρώιμα στάδια οι αρχές ε, είχαν ε, και θέματα επικαλύψεων με τα παλιά προγράμματα και τα καινούρια. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτός ο ρυθμός ε, ε, τους μήνες βελτιώνεται σταθερά. Ε, η απορρόφηση πλησιάζει πλέον ε, τους ρυθμούς του 2013 και όσον αφορά τις υποχρεώσεις που έχουμε στο δεύτερο πίνακα Βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει ε, τα επίπεδα του περίοδου 2007-2013. Είναι σημαντικό να έχουμε τους ρυθμούς πληρωμών όπως τα πληρωμών στα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Βλέπουμε στο τέλος του 2017 και το ποσοστό πληρωμών και βλέπουμε την ισοδύναμη κατάσταση για την περίοδο 2007 με 2013. Η Ολλανδία έχει φτάσει 24% των πιστώσεων Προχωράμε λοιπόν βλέπουμε τα, ε, το για όπου ε, στα κράτη-μέλη ε, αντιπροσπεύει συγκεκριμένα προγράμματα πολιτικής συνοχής και βλέπουμε διαφοροποιήσεις, σημαντικές διαφοροποιήσεις. Το πεδίο εφαρμογής είναι πιο ισχυρό σε κράτη-μέλη που έχουν αποκεντρωμένο σύστημα και που έχουν πολλά προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται. Μπορούμε να βρούμε διάφορες εξηγήσεις για αυτές τις διαφοροποιήσεις γιατί υπάρχουν σημαντικές διαφορές ε, στους ρυθμούς πληρωμών σε χώρες με λιγότερα ε, προγράμματα και πιο ε, συγκεντρωτικό χαρακτήρα. Έχουμε δύο κόντεξτ, ένα εξωτερικό και ένα στο πλαίσιο της ΕΣΥΦ, του ΕΣΥΦ οι παράγοντες από το εξωτερικό πλαίσιο είναι οικονομικοί παράγοντες, όπως είναι ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης, που είναι πολύ σημαντικός. Οι αρχές πραγματικές έχουν ε, θέματα στην εφαρμογή όταν αντιμετωπίζουν ε, τη μετατόπιση των αναγκών εξαιτία της ε, κρίσης και των αλλαγών και την, ε, τις αλλαγές στη διάρθρωση των οικονομικών αγορών. Έχουμε λοιπόν μια καθυστέρηση στην εφαρμογή. Επίσης, σε πολλά κρατημέλη δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για να χρηματοδοτήσουν ε, ε, προγράμματα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια υπάρχει μεγάλη έμφαση στην ποιότητα της διακυβέρνηση στα προγράμματα για την πολιτική συνοχή. Υπάρχουν ρυθμίσεις σε κάθε κράτος μέλη για να υπάρχει αποδοτικότητα, ρυθμιστική ποιότητα κτλ. Υπήρξε ένας διαχωρισμός ε, μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρω... Ε, χωρών Υπάρχει και μια άλλη ομάδα ε, του Νότου και του Βορρά που έχει την υψηλότερη απόδοση. Έχουμε δει πρόοδο από τις ε, χώρες του U12 όπου υπάρχει η χαμηλότερη ποιότητα διακυβέρνησης και παρόλα αυτά ε, μπορούν να πετύχουν καλύτερη απόδοση υπάρχουν ε, διαφοροποιήσεις ε, στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και αυτό είναι κάτι που τονίστηκε στην εκ ε, αξιολόγηση που έγινε το 2013 από την Επιτροπή. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις θετικού spillover όπου η αποδοτικότητα επωφελήθηκε και σε άλλους ε, τομείς ε, όπου ήταν ε, χαμηλή η απόδοση. Δεν υπάρχει ιδανικό πλαίσιο. Αλλά η εφαρμογή και η πολιτική συνοχής πρέπει να βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με το εθνικό πλαίσιο. Μπορεί να βελτιωθεί η εφαρμογή βραχυπρόθεσμα Τέλος, όσον αφορά το εξωτερικό πλαίσιο, πρέπει να δώσουμε έμφαση σε τομείς όπου εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες κρατικές ενισχύσεις, δημόσιες συμβάσεις δημιουργούν ένα μεγάλο ε, περιθώριο λάθος εξαιτία ε, του ψηλού ε, ποσοστού ρύθμισης διαφορετικών ερμηνεών που μπορούν να δοθούν στο πλαίσιο του κάθε κράτους μέλους. Οι συνέπειες των σφαλμάτων από τις δημόσιες συμβάσεις και τις κρατικές ενισχύσεις είναι ε, να υπάρξει απόσυρση, ε, στέρηση χρηματοδότησης ή να ε, επιβληθούν επιπλέον απαιτήσει. Αυτό ουσιαστικά αποθαρρύνει τους δικαιούχους είτε δεν είναι ικανοί να συμμορφωθούν με τους κανόνες και δεν θέλουν να αναλάβουν το ρίσκο και δημιουργεί πρόβλημα στην εφαρμογή των πολιτικών συνοχή και δημιουργεί και αναγκή για περαιτέρω χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω το λόγο στο Φάμπεν για την υπόλοιπη παρουσία. Okay, ευχαριστώ πολύ. Αφού ακούσαμε λοιπόν για τους εξωτερικούς παράγοντες, σας δούμε τώρα το πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και τις καθυστερήσεις. Όταν βλέπουμε τις καθυστερήσεις υπάρχει καταρχάς το θέμα της καθυστέρησης του νομοθετικού πακέτου το οποίο υιοθετήθηκε τελικά λίγες μέρες μόνο πριν από, τα, από την εκκίνηση των λειτουργικών προγραμμάτων. Αυτό οδήγησε επίσης ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να καθυστερήσουν τις εφαρμογές. Βλέπουμε ότι το συνολικό ποσό των απαιτήσεων και όχι κάποιες ε, μεμονωμένες διαδικασίες και κάποιοι μεμονωμένοι κανόνες. Ίσως λοιπόν το σύνολο της διαδικασίας είναι κάτι το οποίο μπορεί να ε, οδηγεί στις καθυστερήσεις. Τώρα βλέποντας τον ε, οικονομικό έλεγχο εδώ και τις ε, ρυθμίσεις οι οποίες ισχύουν για την παρακολούθηση των διαδικασιών βλέπουμε ότι οι ανθρώπινοι πόροι είναι περιορισμένοι και το προσωπικό το οποίο ασχολείται με τις διαδικασίες ε, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα διαθέσιμο για την επιλογή των προγραμμάτων ή για την οργάνωση ε, σημείων ενημέρωσης ε, του κοινού για τις δυνατότητες ε, χρηματοδότησης. Ένα, μια άλλη αιτία για τις καθυστερήσεις είναι οι υποχρεώσεις για την δημιουργία ειδικών εφαρμοστικών μέτρων όπως τα χρηματοδοτικά μέσα ανάπτυξη συγκεκριμένων περιφερειών ή τα λεγόμενα ITI. Όλα τα μέσα αυτά απαιτούν μία μακρόχρονη προγραμματική φάση. Στην ουσία προγραμματίζουμε για τρία χρόνια, αλλά καλούμεθα να το εφαρμόσουμε σε δύο. Υπάρχει λοιπόν και εδώ ένα πρόβλημα. Τα στοιχεία ΕΦΣΗ λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει μια κάποια επιτάχυνση τον τελευταίο καιρό. Τώρα από, τις, ε, από τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας βλέπουμε και άλλους το, ε, λόγους καθυστέρησης όπως το είδος ε, των ποσών καθορίζεται από το ποια γενική διεύθυνση είναι υπεύθυνη και ποια καλύπτει το πεδίο εφαρμογής. Σε συνολικό επίπεδο όμως το τύπος του Ταμείου δεν εξηγεί τα πάντα. Βλέπετε εδώ ότι τα επίπεδα πληρωμών για τα μεμονωμένα ταμεία είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. Ταυτόχρονα και οι περιφερειακές κατανομές σε επίπεδο εδαφικής συνοχής, μιλάμε για τις λεγότερο προχωρημένες περιοχές, για τις προχωρημένες περιοχές και για τις υπομετάβαση περιοχές. Και εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις διότι το περιβάλλον το οικονομικό ποικίλει αλλά και σε συνολικό πάλι επίπεδο δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. By contrast, when we look at the thematic objectives, there's significant difference in the payment rates between the various, the, the 11 thematic objectives. Thematic objective 3. Ο στόχος 3, τώρα οι περιοχές στόχου 3 και οι θεματολογικοί στόχοι 8 πηγαίνουν σχετικά καλά ενώ ταυτόχρονα το ICT στο θεματολογικό στέχο 2 και 4 έχουν αρχίσει να καθυστερούν. Εδώ είμαστε δυστυχώς υποχρεωμένοι να διακόψουμε διότι όπως είπαμε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε υπέρβαση του ωραρίου εργασίας. So there would be new beneficiaries who would need to be familiarized with the rules of procedure of cohesion policy first. Um,